Καλημέρα σας. Αν δεν απατώμε θα αρχίσουμε. Δεν είναι η συνήθις αίθουσα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σας καλωσορίζω όλους στην πρώτη μας συνάντηση της ΙΜΚΟ του 14. Ελπίζω να αναπαυθήκατε δεόντως κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τους βλέπω όλους φρέσκους φρέσκους και ιδίω την πρώτη εισηγήτρια. Δυστυχώς δεν είμαστε στη συνήθι μας αίθουσα και χρειάζομαι κι άλλα για να τους βλέπω όλους. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν όσοι μας κοιτάζουν από το δίκτυο. Αλλά τέλος πάντων όσοι έχουν έρθει τώρα στο Ιντερνετ τους καλωσορίζω και αυτούς. Λοιπόν, πρώτα τα τυπικά. Να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει μια αλλαγούλα στη σειρά των θεμάτων. Δηλαδή μετά την ψηφοφορία Μάντες για την εντολή της πρότασης του κ. Μάντες, ο κ. Σβάμπ θα κάνει την παρουσίασή του για τις τροπολογίες για το θέμα του και μετά θα μιλήσω εγώ για το θέμα μου. Σε λίγο θα ζητήσω ενημέρωση για τα θέματα που συζητούνται στον τριμερή διάλογο. Μία σύντομη παρουσίαση δηλαδή για το θέμα των ήττα τιμολογίων. Λοιπόν, πρώτα είπα τα τυπικά. Φαντάζομαι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σας υπενθυμίζω ότι τα έγγραφα της συνεδρίασης είναι διαθέσιμα και ηλεκτρονικός, διότι θέλουμε να εφαρμόζουμε το paperless office. Θα το ξέρετε, δεν ξέρετε αυτή την έννοια από την περιασμένη συνεδρια συνεδρία 27-28 Νοεμβρίου τα πρακτικά θα εγκριθούν αν δεν ακουστούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Θα το αναλάβει το θέμα αυτό ο Πάνος Κωνσταντόπουλος. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στον τριμερή διάλογο. Η Βαρβάρα Βάιλερ είναι παρούσα όχι. να σας κάνω εγώ μια ενημέρωση εκ μέρους της κυρίας Βάιλε για την οδηγία που συζητιέται στις, από τις 19 Δεκεμβρίου και έχουμε καταλήξει σε πολιτική συμφωνία για τις ραδιοφωνικές ή εγκαταστάσεις ή τα ραντάρ. Ε, έχουν βρεθεί λέει ικανοποιητικές συμβιβαστικές προτάσεις, ας μην υπησέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά αφορούν θέματα όπως το εύρο της οδηγίας, το κατά πόσον πρέπει παντού να καταγράφονται αυτές οι εγκαταστάσεις για να διαπιστώνεται αν υπάρχει παραβίαση των κανονισμών και την ηλεκτρονική σήμανση για μελλοντικά μηχανήματα όπως τα smartphones για να δούμε αν συμφωνούν όλα αυτά με την νομοθεσία. κυρία Βάιλε τα έχει εξετάσει όλα αυτά εξονυχιστικά. Λοιπόν, άλλα δύο συνδεδεμένα θέματα για την εποπτεία της αγοράς και την ασφάλεια των καταναλωτών όπως ξέρετε τελείωσε η σχετική ψηφοφορία και ο εισηγητής μας είναι συνεχώς σε επαφή με την Προεδρία ο κ. Σέλταν Μόζερ να μας ενημερώσει για το πού βρίσκονται αυτές οι συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, πράγματι, δεν υπάρχουν τόσα πολλά καινούρια να σας αναφέρω. Ακόμα περιμένουμε να υπάρξουν οι λύσεις αλλά η ελληνική προεδρία προσπαθεί να πάρει εντολή για διαπραγματεύσεις μαζί μας εργάζονται στο θέμα είχαν συνάντηση χθε, θα έχουν συναντήσεις και σήμερα και προσπαθούν να πάρουν την εντολή την επόμενη εβδομάδα στην Κορεπέρ έχουμε ακόμα κάποια ευκαιρία να καταλήξουμε σε συμφωνία, αν καταλήξουν σε εντολή από πλευρά τους. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως είχε αναφερθεί και πριν από τα Χριστούγεννα, δεν είναι απίθανο να πρέπει να πούμε ότι δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τις κοινοβουλευτικέ διαδικασίες. Και έτσι συμφωνήσαμε τους κοιόδης εισηγητές στο Κοινοβούλιο. Θα έχουμε αυτή τη διπλή στρατηγική που θα ακολουθήσουμε. Επ' αυτής εργαζόμαστε. Να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε διαπραγματεύσεις, αλλά αν δεν τα καταφέρουμε, να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε με την έκθεση στην Ολομέλεια. Και ταυτόχρονα εργαζόμαστε για διαπραγματεύσεις και για την ψήφιση στην Ολομέλεια της έκθεσης όσο το δυνατόν αργότερα δηλαδή σε σχέση με την κοινοβουλευτική μας εντολή Μάρτιο ή Απρίλιο ίσως. Αλλά αυτό σχεδιάζουμε, να καταλήξουμε την έκθεση στην Ολομέλεια, εν πάση περιπτώσει. Θα ξέρουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα. Και είναι κατά το μάλλον ήταν η απριλιο ισως αλλα αυτο σχεδιαζουμε να καταληξουμε την εκθεση στην ολομελεια εν παση περιπτωση θα ευκαιρία που θα έχουμε. Αλλά αναμένουμε ακόμα και ελπίζω ακόμα και εγώ ότι θα καταφέρουν να βρουν συμβιβαστικές προτάσεις και λύσεις. Γνωρίζω, γνωρίζω ότι Υπάρχει προσπάθεια να καταλήξουν σε συμβιβασμούς, να βρεθούν συμβιβασμοί και λύσεις γύρω από το άρθρο 7 την, το περιβόητο αυτό άρθρο. Αναμένουμε λοιπόν, έχουμε μια διτή, διπλή στρατηγική, θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες στην επόμενη συνεδρίαση. Την επόμενη εβδομάδα θα γνωρίζουμε περισσότερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την ενημέρωση. Θα έχουμε και άλλη μια ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε κατά τη συνάντησή μας στα τέλη του, του μηνός, 22-23 του μήνα. Επίσης εφιστώ την προσοχή σας ότι ο Έλληνας Υπουργός Αρμόδιος, ο κύριος Χατζηδάκης, Υπουργός Ανταγωνισμού, όλοι θα θυμούνται ότι ήταν πρώην συνάδελφός μας Ευρωβουλευτής, στις 3 η ώρα, στις 22 Ιανουαρίου θα είναι μαζί μας, θα είναι παρόν στη συνεδρίαση. Γνωρίζω ότι προσωπικά ενδιαφέρεται σε αυτό το χαρτοφυλάκιο και σε σχέση με τα θέματα της ελληνικής προεδρίας και από πλευράς μας ε, και όλοι και οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα, είναι παρόντες και παρούσες και Είμαι βέβαιος ότι η κυρία Σάρντε Μόζε θα μπορέσει να θέσει ερωτήσεις για αυτό το οποίο ελπίζουμε ότι θα σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ως θέμα. Τώρα προχωράμε στο θέμα του invoicing, λογαριασμούς ε, και έχουμε συμφωνήσει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ε, η κυρία Λάγκεν θα λάβει τον λόγο για να μας ενημερώσει. Παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ναι, καλή σας μέρα πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σε όλους σας καλή χρονιά πρώτα απ' όλα. Άμεσα μετά την απόφαση από πλευρά ΣΥΝΚΟ ξεκινήσαμε το χρονοδιάγραμμα με τη γραμματεία να το σχεδιάζουμε και να το προετοιμάζουμε. Υπήρξε χθε μια πρώτη τεχνική συνεδρίαση και προχθές σε επίπεδα εργασίας με τις γραμματείες και τώρα σήμερα θα έχουμε την πρώτη συνάντηση σχεδόν εισηγητών. Και στη συνέχεια θα έχουμε περαιτέρω συναντήσεις στις 15 Ιανουαρίου τον πρώτο τριμερή διάλογο θα έχουμε τεχνική υφή συνεδριάσεις και στις 22 Ιανουαρίου τον δεύτερο τριμερή διάλογο που ελπίζουμε θα καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Τα κύρια σημεία ήδη καταδεικνύεται ποια είναι. Υπάρχουν διαφορετικά σημεία όπου μπορεί να επιληθούν αυτά. Δύσκολο, πολύ δύσκολο θα είναι το θέμα του χρονοδιαγράμματο γιατί τα κράτη-μέλη θέλουν να έχουν μεγαλύτερες προθεσμίες υλοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί και εκείνη να υπάρχουν τέτοιου είδους δυνατότητες ε, προώθησης ε, και δεν ξέρω πώς όλα αυτά θα μπορέσουν να συμβιβαστούν. Πρέπει να αναμείνουμε την πρώτη συνάντηση σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να σημειωθεί πρόοδο. Μια και στο τέλος θα εγκρίνουμε όλο το πακέτο για τι δημόσιε προμήθειε στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Καλό θα ήταν και τα θέματα των λογαριασμών και τη. Ε, ε, αυτού του χαρτοφυλακίου να ολοκληρωθεί. Η ελληνική προεδρία μας πρότεινε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την έκθεση του κυρίου Μάντες για τα οχήματα και μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος. Ελπίζω λοιπόν ότι θα είναι δυνατόν αυτό να προωθηθεί. Προχωράμε λοιπόν στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διαταξής μας ε, για σήμερα όσον αφορά το υποεξέλιξη έργο είναι, η ενία είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ο κύριος Κοφεράτη που είναι εισηγητής για αυτό το θέμα γνωρίζω ότι θα υπάρξει καθυστέρηση από πλευρά συναδέλφου. Θα δώσω τον λόγο πρώτα στους άλλους γεώδεις εισηγητές. Δεν είμαι βέβαιος ποιος για τους φιλελεύθερους ε, θα λάβει τον λόγο. Η κυρία Ρούιλε είναι παρούσα, εγώ είμαι παρόν. Είμαστε αρκετοί για να γίνει η συζήτηση όπως πρέπει για το θέμα της διακυβέρνησης ενιαίας αγοράς και θα δούμε και τις συμβαστικές προτροπολογίες και ποια πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί. Έχετε τον λόγο κύριε Κοφεράτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλή σας χρονιά, συνάδελφοι. Καλώς όρισαν και οι προσκεκλημένοι μας. Πριν από λίγες μέρες σας έστειλα 11 συμβαστικές τροπολογίες. Και θα σας στείλω και άλλες ε, προτάσεις συμβαστικές για κάποια θέματα τα οποία ακόμη ε, κερμούν. Έχουμε αυτές τις 11 λοιπόν ε, συμβαστικές τροπολογίες. Φαντάζομαι δεν είχατε το χρόνο να τις μελετήσετε γιατί δεν θα προλάβατε. Εγώ φταίω. Δεν εσείς που εστάλησαν τόσο αργά αφορούν την έκθεση όσον αφορά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Δεν νομίζω να έχουμε σημαντικά προβλήματα. 1 έως 5 και 11 Επίσης έχετε υποβάλει και εσείς κάποιες τροπολογίες που χωρίς δυσκολία τις κάλυψα. Περιμένω να μου πείτε τη γνώμη σας και θα τη λάβω υπόψη. Τώρα, έχουμε την ε, συμβαστική 4 που αφορά την ενιαία αγορά στον τομέα της ενέργειας. Και είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα προκρατεύσουμε τους πιο ευάλωτους καταναλωτές. Επίσης, κάτι θα πρέπει να πούμε, ώστε να υπάρχει η ικανοποιητική πρόσβαση για όλους τους καταναλωτέ. Μετά έχουμε τη συμβαστική υπαριθμών 6. Εκεί έλαβα υπόψη τις προτάσεις που έκανε ο κύριος Χατζημαρκάκης ο κύριος Κάκης σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη χρηματοδότησή του στην ε, συμβαστική 7. Εδώ Αντικειμενικά πρόκειται για την πιο δύσκολη διάταξη γιατί έχουμε να κάνουμε με την κινητικότητα των εργαζομένων. Έχουμε εδώ κάποιες ε, τροπολογίες που ε, μεταξύ τους διαφέρουν πολύ. Το θέμα είναι δύσκολο και πολύ σημαντικό. Προσπάθησα να καλύψω όλες τις γνώμες. Με αυτές τις τροπολογίες ανάλογα με τις απόψεις που την τελευταία φορά διατυπώθηκαν και να δούμε τι θα γίνει, πρέπει να ισχύσει η ελεύθερη διακίνηση και να έχουμε όλες τις εγγύσεις για αυτά τα δικαιώματα, να έχουμε βέβαια και τις ε, προεκτικές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για αυτούς που θέλουν να μετακινηθούν, τους εργαζομένους. Στις μερικές τροπολογίες 9 και 10 κάλυψα τα όσα είχαν προτείνει ο πρόεδρος Χάρμπορ και ο κύριος Σουάμπ. Εκκρεμούν ακόμη τρία ζητήματα. Όπως προείπα, προσπαθώ να συντάξω σχετικές συμβαστικές προτάσεις. Πρώτα πρώτα έχουμε την παραγραφό 10 για την βιομηχανική πολιτική που νομίζω ότι θα πρέπει ε, κάτι να πούμε πάνω σε αυτό όπως συζητήσαμε και την τελευταία φορά. Και ο πρόεδρος Χάρμπορ και ο συνάδελφοι αναφερθήκανε στο ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιε είναι οι αρμοδιότητέ μα, να μην συγκρουστούμε για τι αρμοδιότητε με άλλε ενωμένε επιτροπέ. Λογικό είναι αυτό, οπότε και εγώ θα προσπαθήσω να βρω μια νέα διατύπωση, θα σα διαβιβάσω όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό το κείμενο, καλύπτοντα τι παρατηρήσει σα και φυσικά και θα καλύψουμε την βιομηχανική πολιτική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχει το κείμενο ισορροπία. Επίσης, παράγραφος 18. Παράγραφος 18 αφορά τη διαδικασία έγκρισης κάποιων νομοθετικών προτάσεων. Ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει για το τι θα πρέπει να εγκρίνεται όσο γίνεται πιο νωρίς, αλλά βέβαια Νομίζω ότι τελικά και εδώ δεν θα υπάρξει δυσκολία και θα τα συμφωνήσουμε. Θα σας στείλω σχετικά σημείωμα. Επίσης έχουμε το 20. Στην παράγραφο 20 έχουμε τις βασικές προτάσεις που προέρχονται από την ε, πράξη για την ενιαία αγορά. σχετίζεται και με την πρώτη παράγραφο που αναφέραμε όσον αφορά την έγκριση των νομοθετικών προτάσεων. Ε, εδώ πέρα έχουμε την ε, μνήμα κάποιων προτεραιοτήτων και επομένω, θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με τη διακυβέρνηση που βέβαια είναι σχετική με το θέμα μας αλλά κάθε αυτή θα πρέπει να προσαρμόζεται στις κάθε φορά προτεραιότητες που συντρέχουν. Οπότε θα πρέπει να έχουμε παράγραφο για τη βιομηχανική πολιτική και επίση άλλη μια παράγραφο όσον αφορά τι προτεραιότητε και το περιεχόμενο τη ε, ενιαία αγορά. Και πρέπει να αναφερθεί κάπου πού πρέπει να προχωρήσουμε όσο γίνεται ταχύτερα σε ποια μέτωπα. Οπότε, αυτά είχα να σας πω. Έχουμε επίσης τι ε, τις 11 συμμετοχές που σας Θα ε, σας στείλω ακόμα μερικές, πάρα πολύ σύντομα και σε ευχαριστώ για τη συνεργασία σας μέχρι τώρα, γιατί νομίζω ότι ε, τα βασικά τα έχουμε θίξει σε αυτό το κείμενο δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να καταβάλουμε μια τελική προσπάθεια. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ κοντά στην ε, διεκπαιρέωση του θέματο. Νομίζω θα υπάρξει γενική συνένεση γύρω από αυτό το κείμενο, γιατί θα καλύψω τι ανησυχίε όλων, ε, όλων των πολιτικών ομάδων που ε, βρίσκονται στην Επιτροπή μα. Στη διάθεσή σα είμαι, αν θέλετε κάτι. Και όποιο θέλει περισσότερη ενημέρωση, προβέβαια, του παράσχω. Μέχρι να έρθει η ώρα της ψηφοφορίας μπορούμε και διμερώς να αναζητήσουμε τις λύσεις που θεωρούμε ότι είναι οι πιο δόκιμες. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Αλλά υπάρχει. Υπάρχει αρκετός χρόνος για να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, και τελικά να δούμε τι θα κάνουμε για να διεκπληρώσουμε αυτά τα θέματα που ακόμα εκκρεμούν. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα κάνατε, ευχαριστούμε πολύ και για αυτές τις συμβαστικές προτάσεις. Νομίζω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ να προχωρήσει η υπόθεση. Τώρα, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Χατζημαρκάκη και να δούμε τι έχει να μας πει από πλευρά των σκιωδών συγκεκριτών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Κοφεράτη επίσης για τις συμβιβαστικές τροπολογίες που προετοίμασε. Γενικά για το θέμα της ε, έκθεσης για την governance, για την λογοδοσία και χρηστή διακυβέρνηση πρέπει να δούμε τι γίνεται για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη αναγνωρίζοντας τις ανισότητες μεταξύ των κρετών των μελών και υποβάλλοντας συγκεκριμένες συστάσεις για το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Θέλω να τονίσω ότι οποιαδήποτε εποπτεία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανεργία των νέων. Και αυτό είναι κάπως το θέμα που απουσιάζει εδώ, η ανεργία των νέων. Συμφωνώ με την ιδέα να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα συμπληρώνουν τις εθνικές πρωτοβουλίες όσον αφορά το επιχειρήν κοινωνικά και να αναλυθεί η μορφή τραπεζών ανάπτυξης με χαμηλό το καδάνια υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να υποστηριχθούν αυτές ιδιαίτερα Πρέπει να ευχαριστήσω για το ότι κάποιες τροπολογίες έλαβαν υπόψη αυτά τα στοιχεία, ιδιαίτερα η τροπολογία για τις ε, αναπτυξιακές τράπεζες. Επίσης ε, καλοδεχούμενη είναι η τροπολογία 10, συμβαστική τροπολογία, όσον αφορά ε, την παραβίαση κοινοτικού δικαίου και τι πρέπει να αναλαμβάνεται ως πρωτοβουλία κατά τέτοιων παραβιάσεων και παραβάσεων. Δεν βλέπω όμως στις συμβαστικές τροπολογίες το θέμα της ανεργίας των νέων να καλύπτεται επαρκώς και όπως θα έπρεπε. Προτάθηκε βέβαια στην τροπολογία 52 κάτι τέτοιο και θα έλεγα ότι θα μπορούσε να καλυφθεί ως προσθήκη στην συμβαστική τροπολογία 8. Μπορούμε να είμαστε φάνταστοι και δημιουργικοί για αυτό το θέμα εκεί, σε αυτό το σημείο. Πρότασή μου είναι να είναι προσθήκη της τροπολογίας, συμβαστικής τροπολογίας 8 αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλε, παρακαλώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Πρέπει να προσθέσω όμως, δεν τις είδα εξειδικευμένα και λεπτομεριακά. Με μια βιαστική ματιά τις είδα. Θα τις δω όμως ε, λεπτομέρειες. Το ερώτημά μου αφορά το θέμα της κινητικότητας και ελεύθερης ε, κυκλοφορίας. Έχουμε εγκρίνει μια οδηγία για την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών ε, πτυχίων και δεξιοτήτων που είναι ένας καλός συμβιβασμός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εδώ σε αυτό το θέμα να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ίσως και εγώ να σημειώσω από πλευράς μου σε σχέση με τα θέματα σχεδόν εισηγητών. Να αναμείνουμε μέχρι και ο κύριος Σουάπ να είναι παρόν ώστε τα θέματα του ΕΛΚ να αναφερθούν όπως πρέπει. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κοφεράτη, διότι οι συμβαστικές του τροπολογίες νομίζω σημαντικά ενισχύουν, ενδυναμώνουν την έκθεση προς την κατεύθυνση που θέλουμε εμείς και να κινηθούμε και έχει μεγάλη σημασία αυτό για για αυτή την κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Σας ευχαριστώ που το κάνατε αυτό. Σε μεγάλο βαθμό το, μεγαλύτερο αριθμό των συμβαστικών τροπολογιών μπορώ να τον υποστηρίξω υποβάλουμε κάποιες προτάσεις ε, επί κάποιων θεμάτων που αφορούν τα ενεργειακά θέματα και τις ενεργειακές υποδομές. Πρέπει να ε, γνωρίζουμε πάντα και να είμαστε προσεκτικοί όταν υποβάλουμε προτάσεις για νέες ε, πρωτοβουλίες. Πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Θα πρέπει να αντανακλάται η σπουδαιότητα της προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών οι κανονισμοί και οι διατάξεις είναι πολύ περίπλοκες γι' αυτό και δεν είναι αναγκαία να καλύπτονται όλα αυτά στο ευρωπαϊκό επίπεδο κατά λεπτό. Σε ευχαριστώ για τη συνεργασία και για την ε, και από πλευρά των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και από μένα με ιδιαίτερη προσοχή να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μεταξύ κρατών μελών για την τιμολόγηση και τις επικοινωνίες. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα πάρουν σάρκα και ε, οστά αυτές οι προτάσεις. Πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις προτάσεις που έχουμε στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Να ενδυναμωθεί η λειτουργία της αγοράς και των εμπλεκόμενων στην αγορά έχουμε ένα σαφές πλαίσιο για την ενθάρρυνση περισσότερης, ε, μεγαλύτερου ανταγωνισμού. Γνωρίζουμε ιστορικά, αν δούμε τα προηγούμενα, ότι οι τιμές ε, για τους ε, καταναλωτές και οι μειώσεις <clears throat> σε σημαντικό βαθμό είχαν τη σπουδαιότητά τους για τους καταναλωτές. Και σε σχέση με αυτά τα οποία ανέφερε και η κυρία Ρούλε και σε σχέση και με τις παρατηρήσεις του κυρίου Χατζημαρκάκη για την ανεργία των νέων, πολύ καλή ιδέα είναι να συνδυαστούν αυτά με αυτόν τον τρόπο. Η συμβαστική τροπολογία 8 είναι, πρέπει να είναι ισχυρή όσον αφορά αυτά τα θέματα. Και θα ήθελα απλά να αναφέρω επίσης ότι έχουμε συμφωνία τη δική μου τροπολογία 41, αρκετά εκτενής τροπολογία για την χρήση αναλυτικών μέσων και εργαλείων ε, για να μετρήσουμε κάποια πράγματα. Θα ήθελα να προτείνω σε σχέση με την τροπολογία για, τους, ε, για την πρόταση αυτή θα ήταν χρήσιμο να βρούμε μια σωστή διατύπωση. Και έτσι λοιπόν για αυτή την καλή συνεργασία, για μια πολύ θετική έκθεση, θέλω να το τονίσω, αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε με θετικό τρόπο. Τώρα, άλλοι συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν. Ο κύριος Βάμπ, μετά η κυρία Γκέπαρτ. Ο κύριος Σβάμπ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγγνώμη που κάπως καθυστέρησα, αλλά παρόλα αυτά θέλω από καρδιάς να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους καλή χρονιά τις συμβαστικές τροπολογίες του συναδέφου Κοφεράτη τις εξέτασα φυσικά με πολύ προσοχή και συνολικά πιστεύω ότι η έκθεση που μας καταθέτει ο κύριος Κοφεράτη και στους συμβιβασμούς ακολουθεί την κατεύθυνση που εμείς πέρυσι ακολουθήσαμε. Μπορεί κανείς ίσως να πει ότι η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης που πέρυσι είχαμε περισσότερο ακόμα βασιζόταν στην αρχική αρμοδιότητα επ' αυτών των θεμάτων πρωτογενός της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και στην αρχική κατεύθυνση του ιδίου του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως ουσιαστικά πιστεύω ότι αυτό δεν αλλάζει τώρα κάτι στο ότι νέα στοιχεία έχουν ε, ενταχθεί. Γνωρίζουμε για το ότι σε τμήμα των εργασιών μας ε, οι ευάλωτοι καταναλωτές είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Τώρα αν αυτό παρουσιάζεται εδώ καλό είναι. Δεν είναι τόσο η στοχοθέτηση της ε, δικής μας κατεύθυνσης για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, αλλά κατ' ουσίαν δεν έχω πρόβλημα με κάτι τέτοιο πρόταση. Το δεύτερο ποιο είναι. Είναι το ότι ίσως θα είχα εδώ μια πρόταση εγώ για την τροπολογία 8 ως συμβιβασμό και σε σχέση με την τροπολογία 27 του Μάκομ Χάρμπορ Προέδρου και της 38 τροπολογίας του κ. Κοφεράτη να συγχωνευθούν μεταξύ τους. Από ό,τι γνωρίζω μία μόνο οδηγία είναι εδώ το θέμα και γι' αυτό έτσι θα πρέπει να τα διατυπώσουμε. Να μην πούμε αυτές οι οδηγίες αλλά αυτή η οδηγία. Είναι μία ας το πω έτσι σταδιακή κλιμακούμενη διαφοροποίηση και ίσως θα μπορούσε κανείς να πει transpose, μεταφερθεί, να μεταφερθεί προς υλοποίηση. Ίσως μπορώ με αυτό να πω ότι είμαι ικανοποιημένος και χαίρομαι γιατί ότι εντάχθηκαν πολλά από αυτά τα οποία είχα προτείνει εγώ, αλλά κυρίως και η σκιώδηση συγγήτρια που δυστυχώς τώρα δεν μπορεί να παραστεί, επειδή στην Οικονομική Επιτροπή λαμβάνει τον λόγο και παρεμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή εκεί. Ένα παρόμοιο θέμα τίθεται για την συμβαστική τροπολογία 5, μπορώ να πω, που πρόκειται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που όπως ξέρετε θέλω να βοηθηθούν με ιδιαίτερο τρόπο. Δεν γνωρίζω απόλυτα τι εννοεί αυτή η τροπολογία Κατά πόσον εδώ δηλαδή εμείς με αυτό το αίτημα, στο δεύτερο τμήμα αυτής της τροπολογίας που λέει strongly supports, ισχυρά υποστηρίζει την πρωτοβουλία να υπάρξει ανάπτυξη ομολόγων, ε, ε, ομο, ε, bonds. Πώς μπορεί κάτι τέτοιο να ενταχθεί χωρίς να ξεπεράσουμε το όριο των αρμοδιοτήτων των δικών μας αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο συνάδελφος Κοφεράτη, ο εισηγητής, ιδιαίτερα με την ετήσια έκθεση μπορεί να δώσει μια σημαντική συνεισφορά για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και ελπίζω αγαπητέ κύριε Κοφεράτη και αγαπητέ κύριε Πρόεδρε Χάμπορ ότι η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου θα εντάξει επαρκώς αυτά τα θέματα. Και αυτό το έργο που επικοδομητικά υλοποιείται εδώ στο τέλος του ευρωπαϊκού εξαμήνου θα αποκτήσει σάρκα και οστά. Εύχομαι στον εισηγητή κάθε επιτυχία από πλευράς μου. Ευχαριστώ. Uh, uh, Εντάξει, σας ευχαριστώ. Άλλη, η κυρία Γκέπαρτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Και από δική μου πλευράς φυσικά τις ε, καλύτερες και θερμότερες ευχές για μια καλή ευτυχή χρονιά για όλους ε, που είναι εδώ παρόντες και παρούσες και να υλοποιηθούν οι επιθυμίες τους όλων. Θέλω τον συνάδελφο μας Σέζιο Κοφεράτη να τον ευχαριστήσω για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε και κάνει και με βάση τις συμβαστικές τροπολογίες. Και πιο πριν αναφέρατε ένα ιδιαίτερο σημείο τον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής και σωστά διαρωτάστε και απορείτε για το ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για να διαγραφεί αυτό το θέμα. Θα ήθελα με κάθε τρόπο κάθετα να πω ότι σφάλμα θα ήταν να απαλληφθεί κάτι τέτοιο. Διότι πρέπει μια ολοκληρωμένη σφαιρική προσέγγιση, ολιστική προσέγγιση να ακολουθήσουμε όπως προτείνει ο κύριος Κοφεράτη. Γι' αυτό το υποστηρίζω όταν λέτε ότι πρέπει να μεριμνήσουμε να σημειωθεί πρόοδος. Θέλω να υπενθυμίσω και κάτι, ότι εμείς σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχουμε συντάξει και μια γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική από πλευρά τη ΕΕ και έτσι και μεγάλη ε, πλειοψηφία. Ήμουνα εισηγήτρια και το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί σήμερα λέγεται ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας αφορά και θα έπρεπε να διαγραφεί, να εξαλειφθεί. Δεν το κατανοώ αυτό. Είναι απόλυτα δυσνόητο. Τώρα, <clears throat> σε σχέση με το κείμενο του κυρίου Κοφεράτη, να διατυπώσουμε τα πράγματα έτσι ώστε να είναι αποδεκτά. Αλλά να διαγράψουμε αυτά τα πράγματα όχι. Θα ήταν σφάλμα, πιστεύω. Και δεν θα μπορούσα να το δεχτώ. Ευχαριστώ. Uh, thank Σας ευχαριστώ. Κανείς άλλος? Κανένας ευρωβουλευτής? Τότε θα καλέσω τον εισηγητή να συνοψίσει και θα θυμίσω μετά το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ και όλους τους σκιώδεις και όλους όσους έλαβαν το λόγο σήμερα και θα ήθελα να σας ζητήσω ιδιαίτερα για θέματα διατύπωσης να μου στείλετε τις παρατηρήσεις σας ηλεκτρονικά γιατί μάλλον έχουμε αρκετό χρόνο για να εξετάσουμε το κείμενο και μπορώ και εγώ να πάρω υπόψη όλα σας τα σχόλια. Τώρα για την ουσία. Το θέμα της ανεργίας των νέων είναι φυσικά πολύ σημαντικό για τον κύριο Χατζημαρκάκη και το υποστηρίζω και εγώ. Η τροπολογία 52 αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα και πρέπει να δω και εγώ με ποιον ποια συμβιβαστική πρόταση μπορώ να τα συνδυάσω όλα καλύτερα. Πρέπει νομίζω να αναφερθούμε συγκεκριμένα σε προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. Είναι τελείως απαραίτητο. Θα βρούμε λοιπόν μια λύση και για την κινητικότητα. Πολύ λεπτό θέμα, το ανέφερε η κυρία Ρούλε. Πρέπει όμως να το βάλω και αυτό στο σωστό μέρος και να βρω την εξισορρόπηση μεταξύ κινητικότητας και δικαιωμάτων των εργαζομένων που κινούνται, που μετακινούνται. Για τον πρόεδρο θα ήθελα, στον πρόεδρο θα ήθελα να πω ότι για το άρθρο 41 είναι μια καλή επαναδιατύπωση και μπορώ να την υποστηρίξω αυτήν που προτείνει. Όσο για την ενέργεια και τις υποδομές της, επίσης συμφωνώ μαζί του. Πρέπει να προσέξουμε να μην γράφουμε πράγματα που μπορεί να παρερμηνευτούν. ανάλογα με τον καιρό και τον τόπο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε εδώ μια καλύτερη διατύπωση για την προστασία των πιο ευάλωτων καταναλωτών χωρίς να δώσουμε λαβή σε τέτοιες παρερμηνίες. Τώρα στον κύριο Βάρμπα, αν μου στείλει και αυτό τις παρατηρήσεις του για τις διατυπώσεις θα του είμαι ευγνώμων. Η παραπομπή αναφορά που βρήκατε στη συμβιβαστική 5 για τα ομόλογα την έχω πάρει λέξη προς λέξη από πρόταση της Κομισιόν και νομίζω ότι είναι πολύ θαραλέο αυτό αλλά όχι δικό μου, δεν είναι δικό μου το θάρρος, είναι θάρρος της Κομισιόν. Καλό είναι να το αφήσουμε ως έχει. Μπορούμε βέβαια να το αποσαφηνίσουμε πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής παραγωγής. Διότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε βιομηχανικά χωρίς αυτές. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα χρηματοδοτήσουμε την καινοτομία και την έρευνα προς όφελός τους. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν τα μέσα να κάνουν έρευνα, αλλά οι μικρομεσαίες πρέπει να στηριχθούν. Σας ευχαριστώ λοιπόν, αναμένω τις περαιτέρω συστάσεις και προτάσεις σας και θα στείλω τις συμβιβαστικές προτάσεις σε όλους μαζί με την αναφορά στη βιομηχανική πολιτική που ζήτησε η Εύελιν. Θα δω λοιπόν πώς θα τα διατυπώσω όλα αυτά αλλά νομίζω ότι ένα από τα κύρια θέματα πρέπει να είναι όντως η βιομηχανική πολιτική, διότι η εσωτερική αγορά και η προστασία των καταναλωτών εξαρτώνται από την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του παραγωγικού τομέα για τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ. πρώτος σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δουλειά σας. Είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξει αυτό σε παξιλά αποτελέσματα. Σας υπενθυμίζω ότι 23 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε την έκθεση. Είναι πέμπτη που θα είναι η επόμενη συνεδριασή μας. Επίσης, έχουμε και άλλες σημερινές συμφορίες την ίδια ημέρα. Οπότε παρακαλώ οι συντονιστές να εξασφαλίσουν ότι όλοι θα είστε εδώ 23 Ιανουαρίου Πέμπτη το πρωί. Δεν θα χρειαστεί να συνδυάσουμε και το απόγευμα, αλλά θα συνδυάσουμε όλο το πρώτο μισό της ημέρας. Η πρότασή μου, πρόταση του κυρίου Σουάμπ, η έκθεσή μας δηλαδή και η έκθεση του κυρίου Κοφεράτη. Uh, Mr. Manders, uh, uh, proposal. Τώρα έχουμε την έκθεση Μάντερς όσον αφορά τα οχήματα. Θα ε, ψηφίσουμε. Ελπίζω έχουμε απαρτία. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάποιοι λείπουν. Φαντάζομαι ο κ. Μάντε έχει κάνει την καταμέτρηση των παρόντων. Πώ αν μπορείτε, βγείτε, ψάξτε στους διαδρόμους και σύρετε εδώ αυτούς που είναι γύρω-γύρω. Για να έχουμε απαρτία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάντερ να μας πει τι γίνεται με τη σημαντική του αυτή η έκθεση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα, να ευχαριστώ όλους. Καλή χρονιά, ε, όλα να πάνε καλά το 2014. Βλέπουμε ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογέ, τόσο περισσότερο λείπουν οι βουλευτέ. Γιατί όλοι έχουν την προεκλογική του εκστρατεία. σε βρω την έκθεσή μου, είδα που κατέληξε κορεμπέρ και δεν μου αρέσει καθόλου. Ακόμα και οι αντίκες ε, είναι αποδεκτές. Και για μένα αυτό είναι σημάδι ότι δεν τους αρέσει μια τέτοια πρόταση. Ούτε καν να γίνει ο κανονισμός δεν θέλουν. Και λέμε τώρα και για τα διασυνοριακά Οπότε ίσως δεν είναι το κατάλληλη στιγμή για να γίνει η τριμερή συνάντηση. Γιατί αφού απέχουν τόσο οι θέσει μα, πού να βρεθεί η συμβαστική λύση. Βέβαια, από την άλλη μεριά, αν δεν δοκιμάσουμε, δεν θα ξέρουμε αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Οπότε, άντε, ναι, α βγούμε στου διαδρόμου, να ψάξουμε συναδέλφου, να έρθουμε εδώ να ψηφίσουν, γιατί χρειαζόμαστε 21. 21. Και τώρα έχουμε μόνο 14 συναδέλφου. Αυτό δεν ξέρω αν έχει κάποιο πληροξούσιο να ψηφίσει για λογαριασμό άλλου. Έχετε εξοδότηση πληροξούσιο. Θέλετε να ψηφίσω για λόγιο Σουάμπ για όλο το ΕΛΚ. Α, ακριβώ, αυτό θέλω να πω. Εκεί το πάω, λέει ο κύριο Μάντα. I want to show that we are willing to find compromise, uh, so for that reason I think it's... Βεβαίως και είμαι πρόθυμος να συνεργαστούμε. Α, καλά, ας γίνει και άτυπο η τριμερή συνάντηση. Και βέβαια, το Συμβούλιο τώρα με την Ελληνική Προεδρία ελπίζουμε ότι θα προτίθεται να περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν να προσεγγίσει τις θέσεις μας. Γιατί τώρα απέχουν πάρα πολλοί θέσεις μας και είναι κρίμα. Να βγω, να βγούμε, να ψάξουμε συναδέλφους. Χάρμπορ, έχω μία πρόταση πιο πρακτική. Μου λέει η γραμματεία ότι το απόγευμα στις 23 του μηνός θα έχουμε την πρώτη ημερήσια. Οπότε μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία μέχρι τότε, μέχρι το πρωί της ίδιας μέρας. Αλλά ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι συμφωνεί με άλλες πολιτικές ομάδες. Αλλιώς δεν θα βρεθούν οι σωστοί ε, ψήφοι που χρειάζονται. Οπότε μας πούν ε, οι συντονιστές τι γίνεται και θα μπορούσαμε επί της αρχής να κάνουμε ε, μια ψηφοφορία για να έχουμε κάποια ένδειξη του πώς πάνε τα πράγματα. Κύριε Γκέμπχαρτ, τι λέτε. Για πέστε μας. Ναι αγαπητέ συνάδελφε, η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα υποστηρίζει την πρόταση του κ. Μάντερς. Έχω μόνο το πρόβλημα ότι δεν ξέρω πού είναι οι συνάδελφοί μου αυτή τη στιγμή. Τηλεφωνούμε αυτή τη στιγμή να τους βρούμε. Ίσως μια άλλη έκθεση να πάρουμε εντωμεταξύ και μετά να έρθουν οι συνάδελφοι και να ψηφίσουμε. Αυτή θα ήταν άλλη δυνατότητα. Όμως ως θέμα αρχής η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα είναι υπέρ της πρότασης του κυρίου Μάντερς. Δεν είναι αρνητική λοιπόν, α το πω έτσι, τοποθέτηση από πλευρά μα. Απλώ για να το διασφαλίσουμε αυτό, επειδή δεν είναι κάποιοι συνάδελφοι παρόντε. Να μην παρεμηνευτεί λοιπόν αυτό. Ευχαριστώ. Ε, the EPP, Mr. Το ΕΛΚ, ο κύριος Σουάμπ και όσον αφορά όλα βαίνουν καλώς με αυτή την έκθεση. Είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Δεν είμαστε όλοι παρόντες δυστυχώς, αλλά είμαστε κάποιοι παρόντες. Μπορούμε να συνεισφέρουμε λοιπόν ώστε να υπάρξει η αναγκαία πλειοψηφία. Όπου το πρόβλημα είναι σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν και εκεί ψηφοφορίες και αυτό είναι μείζον πρόβλημα. Well, uh, I, right, let me, let me, Um... Να σας υποβάλω μια πρόταση λοιπόν και εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής για αυτό το θέμα και επιβεβαιώνω συμφωνώ με αυτά που αναφέρθηκαν. Είναι σαφές θα υπάρξει αυτή η εντολή. Όλοι υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση. Η πρότασή μου λοιπόν επ' αυτού είναι ουσιαστικά αυτή την υιοθέτηση και υποστήριξη από όλες τις ομάδες το θεωρώ σαφή εντολή σε εμά να προετοιμαστούμε όσον αφορά το Συμβούλιο για τις τακτικές διαδικασίες για τον πρώτο τριμερή διάλογο στις 23 το απόγευμα. Πρότασή μου να ψηφίσουμε επίσημα προς επιβεβαίωση αυτής της εντολής το πρωί της 23ης να καταστήσει σαφές προς το Συμβούλιο ότι όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία και δεν αμφισβητείται η εντολή. Και έτσι θα συνεχίσουμε με τις προετοιμασίες γι' αυτό χωρίς να υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα και αυτό σε σχέση με το ε, να ε, βρεθούν οι αναγκαίοι ε, συνάδελφοι με γοργές διαδικασίες για επιβεβαίωση τώρα. Υπάρχει σαφέστατη τοποθέτηση από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Αν συμφωνούν οι άλλοι και οι συντονιστές σε σχέση με αυτά τα οποία πρότεινα, αυτό προτείνω να γίνει και αυτό να υιοθετηθεί. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Συμφωνείτε με αυτό που είπα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω αυτά που είπατε. Είναι η καλύτερη, λύση πιστεύω. Και εγώ θα ήθελα να έχουμε ευκαιρία να ψηφίσουμε στην Ολομέλη για τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Γιατί όπω επεξήγησα, δεν το βλέπω να είναι τόσο εύκολο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να εξευρεθεί συμβιβασμό. Ένα μήνα όλο και όλο για να διαπραγματευτούμε όλα αυτά τα θέματα. Και ο πρώτο τριμερή διάλογο θα είναι στι 21, 21 Ιανουαρίου ε, και τότε νομίζω δύσκολο θα είναι να μπορέσουμε να βρούμε ένα συμβιβασμό στο τέλος. Γι' αυτό το λόγο θέλω να έχουμε μια ευκαιρία στην Ολομέλεια να μπορέσουμε να ψηφίσουμε για το, την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης. Να μην πάει στράφη η δουλειά μας. Ευχαριστώ. Εντάξει, μπορούμε να το εγγράψουμε για το μάτιο ε, στις εργασίες της Ολομέλειας και να υπάρχει και κάποια ελαστικότητα αν προχωρήσουν με ικανοποιητικό ρυθμό οι διαπραγματεύσει, ώστε να έχουμε την τελική ψηφοφορία για αυτό τον Απρίλιο, να επανέλθουμε τον Απρίλιο, να έχουμε άλλο ένα μήνα διαπραγματεύσεων πρωτού ολοκληρωθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο. Να συνεχίσουμε λοιπόν να προετοιμάζουμε τις διαδικασίες ε, για την Ολομέλεια του Μαρτίου και να δούμε και τις δυνατότητες που θα υπάρχουν να ε, προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευελπιστώ ότι θα σημειωθεί πρόοδος αυτό το χαρτοφυλάκιο. Να υπενθυμίσω <clears throat> σε εσά ε, το ότι στις 23 Ιανουαρίου 22 διορθώνει ο πρόεδρος το απόγευμα ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης από την Ελλάδα θα θα είναι παρόν. Μπορείτε να έρθετε να θέσετε ερωτήσεις ε, για τη γραμμή που ακολουθεί και την πρόοδο που σημειώνει η Ελληνική Προεδρία για αυτά τα θέματα. Τρεις η ώρα λοιπόν 22 Ιανουαρίου ο κύριος Χατζηδάκης θα έρθει στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Ελπίζω αθρώα να είναι η συμμετοχή σας ώστε να έχει επιτυχία αυτή η συνάντηση. Ωραία, προχωράμε λοιπόν στη συνέχεια στο επόμενο θέμα που είναι η έκθεση του κυρίου Σβάμπ, σημαντική έκθεση του κυρίου Σβάμπ για την ασφάλεια στο δίκτυο, στο διαδίκτυο, ασφάλεια δικτύων. Έχουμε συμβαστικές τροπολογίες, τρεις που πρέπει να εξετάσουμε σκιώδεις εισηγητές Ραμών, ε, Μάντας παρόντες είσαστε οι γι' αυτό ο κύριος Έγκστρομ απουσιάζει θα έρθει ο κύριος Έγκστρομ τι ξέρετε και εγώ είμαι παρόν ο σκιώδης εντάξει λοιπόν ας προχωρήσουμε καλό τον κύριο Σβάμπα να παρουσιάσει συμβαστικές τροπολογίες Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίως αγαπητοί σκιώδεις εισηγητές πρέπει να πω για τη δυνατότητα που μας δίνεται σήμερα αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες να μπορέσουμε να τις παρουσιάσουμε που εχθές σε μια συνάντηση σκιωδών εισηγητών είχαμε προσυζητήσει ήδη. 232 συνολικά τροπολογίες κατατέθηκαν στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 98 τροπολογίες της αρμόδιας Κοινοβουλικής Επιτροπής ε, επί της ουσίας Ήτρε, όπου η συνάδελφος Πιλάρντερ Καστίγιο εξαιρετική ψήφιση, ψηφοφορία διασφάλισε, ώστε πραγματικά επί της ουσίας και στις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές βρισκόμαστε ενταγμένοι σε μία κοινή κατεύθυνση και γραμμή. Ευχαριστώ γι' αυτό. Και η ΑΦΕΤ τοποθετήθηκε και αναμένουμε την ψήφιση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ, που θα ψηφίσει το θέμα την επόμενη Δευτέρα και από πλευρά ε, εισηγητού της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ υπήρξαν κάποιες διαφορές στην αρχή κάποιες τριβές, ε, ποια σπουδαιότητα έχει η προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων και πώς τα προσωπικά δεδομένα και η προστασία τους θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο. Εργάστηκε και συνεργάστηκε επικοδομητικά η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθεριών ώστε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό όπως αυτό που έχουμε θα ψηφιστεί λοιπόν σε σχέση με την ε, ε, Επιτροπή αυτή στις 13 το θέμα. Πρέπει να αναμείνουμε την ψήφιση. Υπάρχει όμως μεγάλη σύμπτωση απόψεων μεταξύ όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Οι 33 συμβαστικές τροπολογίες που έχουμε μπροστά μας με την τροποποίηση της αλλαγές που συζητήσαμε χτες ανταποκρίνονται σχεδόν ακριβώς σε αυτά που ήθελε να πετύχει η κοινοβουλευτική μας επιτροπή πλειοψηφικά. Αν επιτρέπετε πρόεδρε τα ουσιοδέστερα στοιχεία να αναφέρω που αφορούν τις συμβαστικές τροπολογίες και τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτές. Πρώτα θέλαμε και το έχω αγγλικά μπροστά μου, θέλαμε να έχουμε μια ενδυνάμωση της πτυχής της, α, του, της εχεμήθειας ή της εμπιστευτικότητας σε σχέση με τους εμπλεκόμενους και έναντι των δημοσίων υπηρεσιών. Δεύτερον, θέλουμε από κοινού, και επ' αυτού δεν υπήρξε καμία διαφορά απόψεων, θέλουμε τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων να τα ενισχύσουμε. Και είναι σαφές ότι όταν προσωπικά δεδομένα διαδραματίζουν κάποιο ρόλο, η ρύθμιση προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα, θα έχει δεσπόζοντα ρόλο. Κυρίως για τις υποχρεώσεις που εκείνοι εμπλεκόμενοι στην αγορά και στην οικονομία ε, επομίζονται στο παράτημα 2 για παράδειγμα όπως αναφέρονται και που έχουν ε, αρμοδιότητα για κάποιες υποδομές. Αυτή η σπουδαιότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των δεδομένων αφορά και το άρθρο 9, το 8 αλλά και το άρθρο 13 και 14 επιπλέον. Τρίτον πρόεδρε. Ιδιαίτερα το αίτημα του κυρίου Ραμών, Γαρσές Ραμών λάβαμε υπόψη. Μια ενδυναμωμένη ευρωπαϊκή καινοτομία να αναλυφθεί έτσι η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα της ασφάλειας των δικτύων να προαχθεί ευρωπαϊκά όπως πρέπει. Δεν έχει αυτό ε, τοποθετηθεί όπως ε, θα έπρεπε ακριβώς αν το καταφέρναμε πριν από 20 χρόνια όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές σε σχέση με τις εταιρείες που δημιουργούν το Airbus σήμερα να, είμαστε, να έχουμε ευρωπαϊκή δράση, στον τομέα λοιπόν της επικοινωνίας εξακολουθούμε να ε, εξαρτώμεθα από αμερικανικές εταιρείες και από κινέζικες εταιρείες παρότι αυτή η πτυχή είναι τόσο σημαντική για μας. Γι' αυτό το αίτημα για τις επικοινωνίες του κυρίου Γκαρσέ Ραμών το υποστηρίζω έντονα. Τέταρτον, Πρόεδρε, θέλουμε να διασφαλίσουμε και αυτό αφορά κυρίως τον συμβιβασμό, συμβαστική τροπολογία 8, οι υφιστάμενες υποδομές, οι υφιστάμενες, οι υφιστάμενες ε, επιτηρήσεις ή εποπτείες υποδομών όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων να μπορεί να παραμείνει και να μην έχουμε διπλές επικαλύψεις ή διπλές δράσεις στον τομέα, για παράδειγμα, των όσων σήμερα εποπτεύονται και πρέπει να αναφέρονται και να υποβάλλονται εκθέσεις, να μην έχουμε θεσμούς εποπτείας ή επιτήρησης. Να παραμείνει η εποπτεία, η επιτήρηση ως έχει και να προσθεθούν οι αναγκαίες πρόσθετες δράσεις. Επιπλέον στο άρθρο 9 έχουμε ενδυναμωμένη συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην οικονομία, στους οικονομικούς κύκλους, market operators, τους εμπλεκόμενους στις αγορές. Ήταν και δικό σας αίτημα, Πρόεδρε Χάμπορ. Έχουμε μια διτή προσέγγιση προς τις ε, ε, δομές ε, εποπτείας, αλλά και από, από την εποπτεία στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στην αγορά ώστε να υπάρχει αμφίδρομη δράση επικοινωνίας στην ενημέρωση και πληροφόρηση. Αυτό το πλαίσιο μπορεί να ενισχυθεί και θα πρέπει να ενισχυθεί. Έκτον, στο άρθρο 10 έχουμε ένα σύστημα πρώιμης έγκαιρης προειδοποίησης και μάλιστα χωρίς ε, περιτές καθυστερήσεις, without undue delay, να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις ε, υπό το πνεύμα της ε, διασφάλισης εμπιστευτικότητας Ό,τι συμβαίνει θα πρέπει όμως άμεσα να μπορούν να το δηλώνουν και η δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών να μπορεί να, συνεχί, να ε, προχωρεί όταν υπάρχουν θέματα που αφορούν ε, δημόσιο συμφέρον ή τους πολίτες. Διαφορετικά θα εντάσσονται στα ε, αιτήσεις εκθέσεις. Έβδομον, για το άρθρο 14 όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης και πληροφόρησης. Έχουν προσαρμοστεί τα πράγματα ώστε οι εμπλεκόμενοι στην αγορά και στην οικονομία να εμπλέκονται ενδυναμωμένα σε αυτή τη διαδικασία Πώ Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση και αποτίμηση των πληροφοριών και υπό την εχεμήθεια και την διασφάλιση του απορρίτου. Ε, και έχουμε διασφαλίσει <clears throat> ότι στο παράτημα 2 δεν θα εντάσσονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά, θα υπάρχει εθελοντικό πλαίσιο, εθελούσιος χαρακτήρας, εθελοντικός χαρακτήρας ένταξής του σε σε αυτόν τον κατάλογο. Επίσης το αίτημα της Επιτροπής Ήτρε ελήφθη υπόψη επιχειρήσεις που έχουν ε, ε, ενταχθεί στο χρηματιστήριο και συμμετέχουν στις χρηματιστηριακές ε, συναλλαγές ως καταγεγραμμένες υπηρεσίες εθελοντικά στις ε, εκθέσεις απολογισμού να μπορούν να εκθέτουν τα σχετικά με κυβερνοεπιθέσεις που παρουσιάζονται ή τέτοιες παρεμβάσεις. Εθελοντικά, όχι όλες οι επιχειρήσεις. Κυρίως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ισχύουν για τις εταιρείε ομολόγων ε, και ε, μετοχών. Έχουμε καταργήσει οποιασδήποτε περιττές διαδικασίες. Πρέπει να είμαστε συνεκτικοί όσον αφορά το νομικό πλαίσιο επ' αυτών. Και κάποια άλλα σημεία, το άρθρο 8 για παράδειγμα, για το άρθρο 15 του πλαισίου των ε, οικονομικών ελέγχων audits, αυτή η τροπολογία σε σχέση με το άρθρο 13α μπορεί να ληφθεί υπόψη, όπου τα κράτη-μέλη διατηρούν την αρμοδιότητα να προβλέπουν πρόσθετους οικονομικούς ελέγχους, audits, αν θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο στην επικράτειά τους. Από με την συνάδελφο Σλούτερ είδαμε ότι στη Σουηδία η παραγωγή ε, μαγιάς ε, για παράδειγμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με συγκεκριμένο τρόπο. Μια και όμως ε, η παραγωγή μαγιάς ε, σε όλη την Ευρώπη δεν θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζεται μια και υπάρχουν περισσότεροι παραγωγοί μαγιάς. Πρέπει να δούμε την δυνατότητα σε σχέση την δική τους αξιολόγηση και αποτίμηση να εντάσσονται και αυτοί σε αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρω τώρα πώς ε, ε, ο κύριος ε, Ραμόν Γκαρσέσα από τους σοσιαλιστές τοποθετείται από αυτού του θέματος. Ο κύριος Λούτερ όμως είπε ότι σε ένα δεύτερο παράτημα θα μπορούσε να ενταχθεί η αλυσίδα των τροφικών, διατροφικών προϊόντων, food chain, παράρτημα για αυτές τις χρήσεις. Για το άρθρο 16 για τις προδιαγραφές θέλω μόνο να πω ότι είναι σημαντικό για μας ε, οι ευρωπαϊκές ε, προδιαγραφές να είναι interoperable, δηλαδή διαλειτουργικές, να μπορούν με δεσμευτικό ε, αξιόπιστο τρόπο να είναι διαλειτουργικές. Πρέπει να είναι open standards, ανοιχτές τέτοιες προδιαγραφές. Όμως αυτό δεν μπόρεσε πλήρως να γίνει δεκτό, γιατί το τι είναι ο ορισμός ενός ανοιχτού τέτοιου πλαισίου προσδιοριστικού πλαισίου δεν είναι σαφές. Εδώ το θέμα της διαλειτουργικότητας νομίζω μπορεί να βοηθήσει να επιτευχθεί αυτή, να καλυφθεί αυτή η πτυχή. Κυρώσεις ε, ε, είναι τότε ε, ε, ε, ενδείκνυνται τότε όταν πλημελώς ή εσκεμμένα κάποιοι υδρούν. Και για το δεύτερο στοιχείο που είναι, ε, αφορά τον πυρήνα της πρότασης για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται, συμφωνήσαμε και είπαμε όλες οι υποδομές στον τομέα εφαρμογής θα εντάσσονται όπου πραγματικά οι αρμόδιες επιχειρήσεις μετά από αξιολόγηση καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτές οι υποδομές έχουν κέρια σημασία και πρέπει να είναι resilient, ανθεκτικές. Όμως κάποιες, ε, κάποιους τομείς ε, δεν τους ε, εντάξαμε επειδή μπορεί στις δομές τους ενδεχόμενα να υπάρχουν κάποιες κέρυες υπηρεσίες που παρέχονται. Και με τον κύριο Γκασέ που έθεσε το ζήτημα κατά πόσον εδώ ε, διάβλη επικοινωνίας platform of communications ε, πρέπει να διανοίγονται για, το, για ποιον λόγο δηλαδή θα πρέπει κάποιες υπηρεσίες από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών να εντάσσονται και κάποιες άλλες όχι είναι πάντα κέρια σημασίας ε, όταν αφορούν αυτές οι επικοινωνίες ε, σπουδές παροχές ή μεγάλη σπουδαιότητας παροχές σε διαφοροποίηση με τις μη κέρυες υπηρεσίες και όταν δεν υπάρχει αυτή η σπουδαιότητα, δεν υπάρχει λόγος να ανταποκρίνονται σε αυτό το πλαίσιο αυτές οι εταιρείε. Πρόεδρε, έδωσα μια επισκόπηση συνολικά για το τι συμβαίνει. Είναι όμως πολύ τεχνικά αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την προσφορά αυτών των κατάλογο να τον υποστηρίξουν σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν κάποια θέματα που από πλευράς γραμματείας πρέπει να εξεταστούν με την νομική υπηρεσία και πιστεύω ότι τότε την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να ψηφίσουμε και να εγκρίνουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very Σας κατευχαριστώ για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει. Χαίρομαι που υπάρχει καλή συνεργασία με την Επιτροπή Βιομηχανίας. Γκαρσίας Ραμόν, επόμενος, ως σκιώδης από τους σοσιαλιστάς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Συνέλεφο Σβάμπ για το έργο του και για τον διάλογο που έχει ξεκινήσει και που ελπίζω να έχει θετική κατάληξη. Χθες συναντηθήκαμε οι σκιώδες με τον εισηγητή. Δεν νομίζω ότι επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει τη σημασία αυτής της οδηγίας. λόγω του θεματότης, λόγω του, του λόγω του περιεχομένου που ε, ε, δίνουμε. Οπότε θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες στην ΙΜΚΟ να πετύχουμε να κάνουμε μια αξιόλογη έκθεση, να υπάρξει συνένεση. Δεν νομίζω ότι η προσπάθειά μας ε, αξίζει το λόγο. Επίσης, αυτή η οδηγία αφορά την ασφάλεια των δικτύων. Κάτι πολύ σημαντικό για την οικονομία, τις οικονομικές αλλαγές, το διεθνές εμπόριο, αλλά η ασφάλεια είναι σημαντική και για τις ε, προσωπικές επικοινωνίες. Και για τον ιδιωτικό βίο, και για τον δημόσιο. επικοινωνία και πληροφορίες ε, σήμερα είναι κάτι το οποίο ε, αποκτά αυξανόμενη σημασία. Ε, γι' αυτό λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς θα πρέπει να είμαστε στη θέση να διαμορφώσουμε κάποιες προτάσεις κατανοητές, ακριβείς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε μια αξιόπιστη λύση για το θέμα αυτό που είναι η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Ακριβώς είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουμε 30 ε, τροπολογίες. Κάποιες από αυτές τις ε, κάλυψε με σημαντικές προτάσεις ο κ. Σουάμπ. Συμφωνούμε επίσης για την πρόταση των ερευνητικών κέντρων, των πανεπιστημιακών κέντρων που θα βοηθήσουν στο να πετύχει η οδηγία τους στόχους της. Επίσης, θεωρούμε ότι σωστά προσέχει η οδηγία το θέμα της διαφάνειας, τα θέματα της ε, κατανόησης των νέων ε, τεχνολογιών που δεν θα πρέπει να αποτελούν φραγμό ε, στο να αισθάνεται ο Ευρωπαίος για όλες τις ε, επαφές για τη χρήση των δικτύων ασφαλής. Χθες συζητήσαμε οι σκιοδοσηγητές το θέμα και ετώνησα ότι δεν θα πρέπει η οδηγία να αφήσει περιθώρια για παρερμηνίες όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην πληροφορία και στην ενημέρωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του περιεχομένου της ε, οδηγίας. Είναι κάτι το οποίο ε, πάρα πολύ επίκαιρο επίσης τη, ε, τη σημερινή Οπότε και είπα ο εισηγητής ότι θα προσπαθήσει να καλύψει αυτή μου την ε, πρόταση. Επίσης, έχουμε κάποια τροπολογία για να καλύψουμε όχι μόνο τα δίκτυα αλλά και τα tablets και τα κινητά και όχι μόνο τους υπολογιστές. Εν κατακλείδη πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε το ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες σε αυτό το μέτωπο ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να μπορούν να επέμβουν κάθε φορά που έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό και έτσι να υπάρχει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη ε, προς τα δίκτυα και τις πληροφορίες. Αυτά, αυτό το χαρακτηριστικό ε, χαρακτηρίζει το ένα κράτος δικαίου από το οποίο θα πρέπει να απομακρυνθούμε ούτε πόντο. Επίσης θα πρέπει να καλύψουμε και τις υπηρεσίες ε, που περιέχονται στο δεύτερο παράδειγμα όσον αφορά τα μηνύματα, όσον αφορά ε, τα δίκτυα διακίνησης, διανομής που αφορούν κυρίως τα ε, γεωργικά και τα διατροφής. Γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με την ε, γεωργία και τη διατροφή. Γιατί αφορούν τη δημοσία υγεία. Είναι ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά για τον κόσμο. Αλλά επίσης και υπηρεσίες διαβίβασης ε, μηνυμάτων, χαρακτηρίζω χαρακτηρίζονται πολλές πλατφόρμες, ε, πολλά, είδη διάβλων τεχνολογικών. Αυτά σχετίζονται με το ζήτημα τη ασφαλής δικτύων ε, που μας απασχολεί και πρέπει να το προσέξουμε. Αυτές είναι οι θέσεις μας και σας ευχαριστώ, προέδρο. Εμεί ευχαριστούμε. Κύριε Μάντε, για το λογο <laughs> ζητώ ε, συγγνώμη που σηκώθηκα και έφυγα, αλλά η τηλεόραση ε, ήρθαν τότε κάποια κανάλια και θέλω να κάνω κάτι δηλώσεις για το θέμα μας. Τέλος πάντων, ευχαριστήσω τον ε, Ανδρέα Σφάμπ και ζητώ συγγνώμη που δεν μπορούσα να έρθω στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών, αλλά πάντως νομίζω ότι το έργο του προσπάθησε να καλύψει τις περισσότερες από τις τροπολογίες. Θα ήθελα να μου πούν οι συνάδελφοι της Άλντε ε, εάν συμφωνούν, αλλά βασικά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε και στην ε, επόμενη συνάντηση των σχεδόν συγκεκριτών που νομίζω είναι την επόμενη εβδομάδα, φαντάζομαι θα τα βρούμε. Οπότε είμαστε σε καλό σημείο, συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα καλά. Okay. Um, I think Κύριε Engstrom δεν είναι εδώ, οπότε να σας πω εγώ μερικά πράγματα. Γιατί ξέρετε, ε, πάρα πολύ προσεκτικοί ήμασταν όσον αφορά την υποβολή τροπολογιών από την πλευρά της δικής μας πολιτικής ομάδας. Πάντως σημειώθηκε πρόοδος. Έχουμε και κάποιες προτάσεις μας σε συμβαστικές που δεν καλύφθηκαν. Αφορούν το πόσο εμπιστευτικό χαρακτήρα έχουν κάποιες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά ε, τα ευάλωτα σημεία των δικτύων. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε θα πρέπει κάποια στιγμή να τηρείται αυτή η μυστευτικότητα γιατί δεν μπορεί να δημοσιοποιηθούν αυτά τα σημεία που σας προανέφερα. Και έχουμε επίσης ε, κάποια σημαντικά σημεία όπως την Ιταλική 28 που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να έχουμε ε, διαβίωση πληροφοριών μέσω ασφαλών δικτύων, ε, αξιόπιστων, να διακρίνεται αυτό από εμπιστευτικό χαρακτήρα. και ότι θα πρέπει οι αρχές να επαγρυπνούν ούτως ώστε ε, να έχουν πιστευτικό χαρακτήρα οι πληροφορίες σχετικέ με τα παρόντα σημεριών δικτύων. Κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον σε μια συμβασική τροπολογία του κυρίου Σουβάμπ έχουμε διατύπωση που δεν ε, συνάδει τόσο πολύ με αυτά τα οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Νομίζω συμφωνεί ο κύριος Βάμπ. Οπότε και εμείς θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ακόμη περισσότερο με τα όσα προτείνει ο κύριος Σουάμπ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Αν συμφωνείτε κύριε Σουάμπ, ε, να δώσουμε το λόγο σε, όποιον θέλει ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα δώσω το λόγο σε εσά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, έχετε διαδεχθεί τον συνάδελφο με τον είχαμε συνεργαστεί, ο οποίος ε, ανέλαβε νέα καθήκοντα. Οπότε πέστε μαζί εσείς τι λέτε και κατόπιν να δώσω το στον κύριο Σουάμπ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που μας υποστήριξε τόσο πολύ σε αυτό το θέμα καθώς και τον εισηγητή κύριο Σβάμπ για την αποτελεσματικότητα και ταχύτητα της εργασίας του. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για επίτευξη συμφωνίας. Γενικά οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και περιγραφεί συνοπτικά δεν αντιπροσωπεύουν καμία ιδιαίτερη δυσκολία για μας εκτός από μερικές λεπτομέρειες. Αναγνωρίζουμε βέβαια, από, αναγνωρίσαμε από την αρχή ότι μόνο αν υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και μεταξύ των κρατών μελών πρόκειται να πετύχουν όλα αυτά καθώς και αν υπάρξει αμοιβαία πληροφόρηση οι δημόσιες αρχές και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να συνεννοηθούν επ' αυτού. Επίσης ανέκαθεν λέγαμε ότι υπάρχουσες δομές σε εθνικό επίπεδο πρέπει να διατηρηθούν και η πολυεπίπεδη δομή που έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα δεν χρειάζεται να επιβαρυνθεί με πρόσθετες δομές. Το μόνο που λέμε είναι ότι το Εθνικό Σημείο Επαφής πρέπει να υπάρχει για να μπορούμε και εμείς να έχουμε ένα συνομιλητή επίσημο. Επίσης σημειώνουμε ότι δεν θα έπρεπε υπερβολικά νωρίς να δίνονται, να χορηγούνται πληροφορίες στο κοινό με τρόπο που να μπορεί να βλάψει τους παράγοντες της αγοράς. Μόνο αν είναι προς το συμφέρον, αν είναι προς το δημόσιο συμφέρον θα γίνονται αυτές οι αποκαλύψεις προς τους ενδιαφερόμενους. Επίσης σημειώσαμε ότι η βιομηχανική και εμπορική διάσταση δεν έχει αγνοηθεί συμπεριλαμβανομένης και της καινοτομίας. Τα ερευνητικά προγράμματα και η στρατηγική είναι κάτι που χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε ότι συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση Ένα μόνο θέμα θέλουμε να θίξουμε. Πώς θα καλύπτονται όλα αυτά. Καταρχήν η δημόσια διοίκηση χρησιμοποιεί όρο και λιγότερα χαρτιά και λειτουργεί ηλεκτρονικά. Επομένως πρέπει και αυτό να καλυφθεί. Επίσης ο ορισμός του ποιοι παράγοντες της αγοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Οι βασικές εταιρείες ίντερνετ που χορηγούν υπηρεσίες πρέπει και αυτές να συμπεριληφθούν. Δεν θέλουμε να υπάρξει περιοριστικό στενός ορισμός του ποιε ηλεκτρονικές υπηρεσίες ακριβώς πρέπει να συμπεριληφθούν γιατί σε 4-5 χρόνια θα έχει αλλάξει το σκηνικό. Και όπως είδαμε και για τα, τις τηλεπικοινωνίες, είναι πραγματική αυτή η ταχύτατη αλλαγή. Παραδείγματος χάρη ανακοινώθηκε ότι η επόμενη γενιά του πιο διαδεδομένου λειτουργικού συστήματος θα βασίζεται αποκλειστικά στο cloud. Θα πρέπει δηλαδή όλοι να συνδέονται σε κάποιο cloud που θα βασίζεται στο Redmond. Εμείς θέλουμε να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελαστικότητα και ευελιξία ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία όλων των βασικών υπηρεσιών κυρίως αυτών που είναι βασικές για την οικονομία μας. Καταλήγω λοιπόν ότι είμαστε αρκετά πολύ ικανοποιημένοι και από την υποστήριξη από την Επιτροπή σας και είμαστε βέβαιοι ότι οποιασδήποτε διαφορές υπάρχουν θα μπορέσουν να επιληθούν και να συμφωνηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σβάμ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συνολικά νομίζω δεν υπάρχουν πολλά στα οποία θα πρέπει να επανέλθουμε. Ίσως άμεσα να συνεχίσω σε αυτό που μόλις είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο τομέας ε, της ε, δημόσιας διοίκησης όπως το βλέπω εγώ, είναι η φύση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης από την οποία απορρέει η υποχρέωση την ανθεκτικότητα των συστημάτων της να την διασφαλίζει. Μεγάλη εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη πρέπει να υφίσταται και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα κράτη-μέλη και χωρίς νομική εντολή εδώ αυτή την υποχρέωση σε κάθε, με κάθε τρόπο θα πρέπει να την λαμβάνουν υπόψη και να ανταποκρίνονται. Αν υπάρχουν αμφιβολίες από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν επικοδομητικό να μας επεξηγούσαν πού τα κράτη-μέλη, σε ποιο σημείο τις υποχρεώσεις για αυτή την ανθεκτικότητα και αντοχή και αξιοπιστία δεν τις διασφαλίζουν για να τα ξαναδούμε. Και σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές ούτε στην Ήτρε ούτε στην Λίμπε δέχτηκαν αυτές τις, ε, ε, αυτά τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν υπάρχουν αμφιβολίες πρέπει να αναφέρεται ποια κρατη σε ποιο σημείο αυτό δεν το λαμβάνουν επαρκώς υπόψη. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο τότε φυσικά θα ήταν κάτι απαράδεκτο και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και θα αντιμετώπιζε την ενιαία αντίσταση της Ευρωβουλής. Όπως όμως επεξήγησα υποθέτω ότι τα κράτη-μέλη θα κάνουν τη δουλειά τους σωστά και θα είναι συνεπή. Τώρα, θα ήθελα, αν γίνεται, σύντομα να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρος όσον αφορά το εμπιστευτικό των ε, ε, δεδομένων αυτών. Αυτή τη συμβαστική τροπολογία ευχαρίστως να την επαναδιατυπώσουμε κάπως. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε σημαντικό βαθμό δεχθεί τη συμβαστική τροπολογία της Ήτρε. Αυτός είναι ο λόγος αυτών των διατυπώσεων που έγιναν δεκτές. Και τέλος, θα ήθελα ένα σημείο να αναφέρω που όπως πιστεύω, όπως θεωρώ, αυτό το χαρτοφυλάκιο το θέτει στο επίπεδο των επίκαιρων συζητήσεων με την αξιολόγηση δεδομένων όσον αφορά τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Διότι αν φυσικά σε όλους είναι σαφές ότι η ασφάλεια των δικτύων είναι υπόθεση των παρόχων αυτών των ίδιων δικτύων, τότε στο ίδιο αυτό το χαρτοφυλάκιο συμβαίνει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε οι πάροχοι που στο μέλλον θέλουν να διασφαλίσουν βελτίωση στο πλαίσιο της ασφάλειας των δικτύων τους, πρέπει να είναι βέβαιοι οι πάροχοι ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζουν στη δημόσια διοίκηση δεν θα τύχουν κατάχρηση. Και γι' αυτό στο άρθρο 6 αποσαφηνίζεται αυτό. Θα μπορούσε να υπάρξει κάποια δυσκολία δυσκολία από πλευρά κάποιων κρατών μελών. Γι' αυτό διασφαλίσαμε με κάθε τρόπο ότι χρειαζόμαστε μία ρύθμιση. Έχουμε ε, τις ε, υπηρεσίες πληροφοριών, ε, έχουμε όμως και άλλα, άλλα δύο θεσμικά όργανα. Δικαστικές ή ε, αστυνομικές αρχές που διώκουν το κυβερνοέγκλημα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ένα τρίτο θεσμό πολιτικού χαρακτήρα που έχουν τα κράτη-μέλη που υπό το πρίσμα της εμπιστευτικότητας και με τους ε, ε, οικονομικά εμπλεκόμενους ε, πρέπει να αξιολογείται ποιοι κίνδυνοι απορρέουν και να αναλαμβάνετε δράση η σύγχυση όλων αυτών των αρμοδιοτήτων μεταξύ κάποιων θεσμών, κρατικών θεσμών ή άλλων θεσμών δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιτρέπεται. Γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη που αναλαμβάνουν τέτοιες αρμοδιότητες και έχουν κάποιες δυσκολίες όπως είναι φυσικό να τα υλοποιήσουν μπορούμε όμως να βασιστούμε από πλευράς Ευρωβουλής ότι όσον αφορά εμάς πρέπει να υπάρχει σαφής ε, διαχωρισμός μεταξύ δραστηριοτήτων μυστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφοριών, της ε, διασφάλισης ε, κινδύνων όσον αφορά την, το έγκλημα και θα χαιρόμουν αν όλοι μπορούσαν να υποστηρίξουν το άρθρο 6 με αυτή τη μορφή. Συμφωνούμε όλοι κατά τα άλλα ότι η ψήφιση την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να απλουστευτεί και να προχωρήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για το έργο που επιτελέσατε. Επιβεβαιώνω ότι θα ψηφίσουμε την επόμενη Πέμπτη. Θα είναι μεγάλη μέρα ψηφοφοριών για αυτές τις ε, μεγάλες εμβέλειας προτάσεις ε, και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτό. Και τώρα προχωρούμε στη δική μου έκθεση, στη δική μου γνωμοδότηση προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεταρρυθμίσεις στο πακέτο τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε να υπάρχει η σωστή διασύνδεση. διασύνδεση. Τον Άντωνη Βίλαν τον καλωσορίζω και σε σχέση με το ποιοι είναι σκιώδεις και είναι παρόντες να διασφαλίσουμε ποιοι θα είναι παρόντες και η κυρία Τόνεν εκπροσωπεί την κυρία Μπάστος δεν ξέρουμε αν ο συνάδελφος ε, θα προσέθει. Θα, θα έρθει ο συνάδελφος. Εντάξει, ο κύριος Κρότσμαν θα προσέθει και αυτός. Τι να κάνουμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα πέντε λεπτών για καφέ, για να προσέθουν. Εντάξει, μια και πρόκειται κάποιοι να έρθουν στην αίθουσα. Ο κύριος Άινστρομ δεν είμαι βέβαιος, μια και απουσίαζε αν θα μπορέσει να προσέλθει ή όχι. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα πέντε λεπτών. Εντάξει, Λοιπόν, ε, υπάρχουν και συσκευές για καφέ έξω υψηλής τεχνολογίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ε, μετά τις ε, και μισή. Στις Ευχαριστώ. her name. Ladies and gentlemen, I think um, I think we have a, a full cast now, so I think. Εντάξει, ήρθαν όλοι. Θα συνεχίσουμε. Καλό θα ήταν να συνεχίσαμε. Βίξτρομ εδώ την είδα. ο κύριε Γκάλλο. Βανχέρν. Τούν. Okay, I think we should make a start, um, if you're happy. Um, so, um... Λοιπόν, καταρχάς Ευχαριστώ τους συναδέλφους που μου έστειλαν ιδέες και βελτίωσαν την έκθεσή μου. Όπως ξέρετε, προσθέθηκαν 300 τροπολογίες και για να σας ενημερώσω που βρίσκομαι. Ευχαριστώ και τη γραμματεία μας που εργάστηκε σκληρά κατά την εβδομάδα των Χριστουγέννων και καταλήξαμε σε 33 συμβιβαστικές. 12, 12. Με συγχωρείτε, αυτό ήταν για την έκθεση ΣΒΑΜ. 12 λοιπόν συμβιβαστικές τροπολογίες για θέματα προστασίας καταναλωτών. Και για να συνοψίσω λοιπόν τα πράγματα, συμφωνήσαμε μεταξύ πολιτικών ομάδων να αλλάξουμε τη δομή της πρότασης της Κομισιόν ώστε τις προτάσεις μας να τις ε, προσθέσουμε για την προστασία των καταναλωτών στην Γενική Οδηγία για τις Υπηρεσίες και νομίζω ότι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμφώνησαν και ελπίζω να μην έχουμε και εδώ προβλήματα γιατί είμαι πεπισμένος ότι πρόκειται για το σωστότερο δρόμο. Τώρα, με τις συμβιβαστικές τι κάναμε. Θελήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις αρχικές τροπολογίες. Δεν τις δέχτηκα όλες όλες τις ιδέες των συναδέλφων, αλλά θελήσαμε να κάναμε μια πολύ επικοδομητική δίωρη συζήτηση Σας ανακοινώνω λοιπόν ότι θα υπάρξει και μια δεύτερη εκδοχή των συμβιβαστικών που θα δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα και θα συμπεριλαμβάνουν τις αλλαγές που δέχτηκα με τους σκιώδεις εχθές. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να σας πω γενικά μόνο τι συμβαίνει. Όλοι οι συνάδελφοι που κατέθεσαν, προτάσαν την κυρία Γκάλο, την κυρία Αρίας, πήραν αντίγραφα και των συμβιβαστικών. Να σας πω λοιπόν μερικές από τις λεπτομέρειες. Ακολουθεί τη δομή και της αρχικής πρότασης η παρουσίαση που θα κάνω. Λοιπόν, καταρχάς υπάρχουν πρόσθετα αιτήματα για περισσότερη πληροφόρηση πριν την υπογραφή των συμβολέων. Εδώ οι αλλαγές είναι ευρέως δεκτές Υπάρχουν και μερικά, μερικές λεπτομέρειες ως προς τις εγκαταστάσεις τερματικών και πώς θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στη νέα δομή των υπηρεσιών και αν αυτό σημαίνει πρόσθετο κόστος πώς θα το διαχειριστούμε. Υπάρχει ένα πιο σημαντικό θέμα πρέπει να το δούμε και στα πλαίσια της δουλειάς μας για τα δικαιώματα των καταναλωτών ευρύτερα που αφορά την εναρμόνιση σε περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζονται τα συμβόλαια που υπογράφηκαν με καταναλωτές. Τη δυνατότητα δηλαδή των καταναλωτών να σταματήσουν να κόψουν ένα συμβόλαιο εάν δεν χορηγείται η υπηρεσία σύμφωνα με τις προσδοκίες τους, δηλαδή ως προς την ποιότητα, την ταχύτητα ή την αξιοπιστία. Θελήσαμε παραδείγματος χάρη να είναι πιο γνωστές οι πραγματικές ταχύτητες που εφαρμόζονται στην ηλεκτρονική επικοινωνία. Αλλά είναι δύσκολο να υπάρξει εναρμονισμένη λύση για όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε ζητήσει και νομική συμβουλή γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα ως προς το πώς σχετίζεται η πρόταση αυτή με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών κυρίως. Πιο λεπτομερείς αλλαγές θα κάνω μετά από τη συνεννόηση με όλους τους κοιόδης, ιδιαίτερα για την περιγραφή του τι αναφέρουν τα συμβόλαια για τις ταχύτητες. Χρειάζεται και αρχική πληροφόρηση και συνεχής πληροφόρηση για την πραγματική χρήση. Υπάρχουν βέβαια τόσο πολλές νέες προτάσεις για τον καθορισμό του τι είναι η βασική ταχύτητα όσο και οι συντάκτες τους. Αυτό που συμφωνήσαμε ως συμβιβασμό είναι ότι για σταθερές συνδέσεις λέει ότι η κανονική ταχύτητα, η ελάχιστη ταχύτητα πρέπει να είναι γνωστή, αλλά για κινητές διασυνδέσεις είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα του δικτύου. Αυτή, αυτός είναι ο συμβιβασμός που βρήκαμε. Συζητήσαμε διαμακρού τις λεγόμενες bundled services, τις συνδυασμένες υπηρεσίες, γιατί είχαμε πει ότι η οδηγία για τις καθολικές υπηρεσίες και τα δικαιώματα των καταναλωτών εφαρμόζονται μόνο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και όχι στις τηλεοπτικές και άλλες ε, πολυμέσων. Υπάρχουν όμως και συμβόλαια συνδυασμένων υπηρεσιών που τις συμπεριλαμβάνουν και άρα το θέμα τίθεται τι, πώς θα διευθετήσουμε ένα τμήμα μιας συνδυασμένης προσφερόμενης υπηρεσίας. Δεν γίνεται μου φαίνεται να εφαρμοστούν οι αλλαγές που προτείνουμε για τα συμβόλαια για αυτές τις συνδυασμένες υπηρεσίες. Αλλά θα το ξαναδούμε αυτό και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να μου δώσει κάποια περισσότερη, πιο εμπεριστατωμένη νομική συμβουλή. Τώρα για τον έλεγχο της κατανάλωσης. Εδώ υπάρχει μια βασική συμφωνία. Συμφώνησα να δεχτώ όλες τις προτάσεις των σκιωδών για τις πήγουσες ή κατεπήγουσες υπηρεσίες που δεν υπήρχαν στην αρχική πρόταση της Κομισιόν και με αυτή την ευκαιρία που είχαμε θελήσαμε να τη συμπεριλάβουμε. Να μπορεί κανείς δηλαδή να συζητήσει και το θέμα αυτό για να προσθεθούν, να ενδυναμωθούν ορισμένες από τις ισχύουσες διατάξεις. κυρία Βανκού ας πούμε, αν και ίσως νέρωσα κάπως τις προτάσεις της, τη συμπεριέλαβα, θα το δείτε. Επίσης τη ζήτησα να αποσαφηνίσει την αρχική της πρόταση για ένα καινούριο 26α Βασικά συμφωνώ, αλλά θα ήθελα περισσότερες αποσαφηνίσεις και την καλό να τις παρουσιάσει. Και τέλος για τη διευκόλυνση της αλλαγής προμηθευτού. Προσωπικά εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να το κάνουμε πολύπλοκο, το θέμα πιο πολύπλοκο από ό,τι είναι, αλλά διαφώνησαν οι περισσότεροι και γι' αυτό τελικά θέλω να είμαστε πιο περιγραφικοί, δηλαδή αυτά που λέει η πρότασή μου που επαναλαμβάνει απλώς την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν για όλα αυτά Ελπίζω να έχετε ικανοποιηθεί από τον τρόπο που χειρίστηκα τις τροπολογίες. Κλείνω λέγοντας ότι το δεύτερο σημείο κλειδί της πρότασης είναι κάτι που αφορά την ανοιχτή πρόσβαση στο ίντερνετ. Και αυτό νομίζω είναι σωστή προσέγγιση. Είμαι υπέρ της διευθέτησης και αυτού του θέματος. Και οπότε έτσι θα εξασφαλιστεί ότι έχουμε ένα συνεπές, ένα ε, στεγανό νομικό πλαίσιο. Έχουμε σχετικά ε, λίγες διατάξεις στον κανονισμό. Και τροπολογίες όμως για την διατύπωση έχω λάβει πάρα πολλές. Τις εξήτασα με μεγάλη προσοχή και οι σκιώδεις συζητητές, όλοι, όλοι όσοι υπέβαλαν τροπολογίες πρόκειται να ε, λάβουμε την απάντησή τους την επόμενη εβδομάδα και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια συνάντηση των σχεδόν εισηγητών την Τετάρτη το απόγευμα ε, οπότε να μπορέσουμε στις 3 η ώρα να συναντηθούμε και με τον κύριο Μπαρνιέ έχουμε μια συνάντηση έχουμε και μια συνέντευξη τύπου να σας πω τώρα για την προσέγγιση δύο λόγια είχαμε από την Μπέρκ με ένα ενημερωτικό σημείο Πάρα πολύ με βοήθησε και έχει φωτίσει πολλά σχολεία σημεία των τροπολογιών. Αυτό το σημείο του Μπέρκ. Κύριε Χάρτα, σας στείλει ένα αντίγραφο, αν θέλετε. Και, κατά γνώμη το ζήτημα ποιο είναι. Ότι Θέλουμε να είναι σαφής η νομοθεσία, να υπάρχει ε, ασφαλεία δικαίου, να μπορούμε εν να έχουμε ως βάση αυτό το νομοθέτημα. Και γι' αυτό ήμουν πάρα πολύ προσεκτικό για κάποιες έννοιες που θα μπορούσαν να είναι δυσνόητες. Best effort, internet. Και αυτό είναι μια τέτοια έννοια. Δεν θεωρώ ότι είναι σαφής, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να περιληφθεί ε, στην ε, έκθεση, στον κανονισμό. Επίσης, εξειδικευμένες υπηρεσίες. Ποιες είναι. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο διαφοροποιεί μια τέτοια εξειδικευμένη υπηρεσία από μια υπηρεσία πρόσβαση στο Ιντερνετ. Γιατί θα πρέπει να έχουμε μια κλινική, μια ξεκάθαρη προσέγγιση. Να υπάρχουν σαφείς διαφορετικές γραμμές και να μην έχουμε κανένα είδους ε, σύγχυση. Απάξι λοιπόν και έχουμε ξεκάθαρους ορισμούς για αυτές τις έννοιες σας που ανέφερα που δεν είναι τόσο σαφείς, τότε θα δούμε πώς θα έρθουν οι τυχόν αντιφάσεις, οι τυχόν α, ε, ε, διαφορές που υπάρχουν και ήδη όσον αφορά κάποια, ε, κάποιες περιπτώσεις δυσμενούς διακρίσεως θα μπορούσαμε να άρουμε αυτή την κατάσταση ε, όλα αυτά τα οποία κάνουν οι κανονιστικές, οι ρυθμιστικές αρχές. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι το οποίο ήδη ισχύει και λειτουργεί και αποδίδει. Οπότε μετά από αυτούς τους σαφείς ορισμούς, είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια αυτές οι εξειδικημένες υπηρεσίες δεν είναι δυνατόν να οδηγούν στην επιδείνωση, στην χειροτέρευση της καταστάσεως, ε, της ευκολίας, αν θέλετε, προσβασιμότητας στο διαδίκτυο. Άρθρο 23, παράγραφος 5. Έχουμε μια τροπολογία της κυρίας Δελκαστήγιο. Ε, σε αυτή τη φάση δεν θα προτείνω συμβατικές τροπολογίες, θα περιμένουμε να δω τι θα βγει, τι θα προκύψει, πώς θα διαμορφωθεί άποψη της κυρίας Δελκαστήγιο. που άλλωστε ε, εργάζεται για την κυρίως αρμόδια επιτροπή, δεν έχουμε κάποια ένσταση σε σχέση με την αρμοδιότητα αυτή. Συγχωρήστε με που μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Οπότε τώρα δώσω το λόγο στους συναδέλφους και όλους και σε όποιον άλλο θέλει να μιλήσει. Κυρία Τούν, για εργασμό κυρία Μπάστος, τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ. Να σας διαβάσω το σημείο που έστειλε η κυρία Μπάστος. Δυστυχώ επειδή θα πρέπει να παραστώ στην Επιτροπή Απασχόληση σε μια ακρόαση για το ρόλο της Τρόικα στις χώρες της κρίσης δεν μπορώ να έρθω στη συνεδρίαση και θα ήθελα πρώτα πρώτα να τονίσω το ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογο το έγγραφο του σχεδίου έκθεσης. Το ΕΛΚ συμφωνεί, Πρόεδρε. Συμφωνούμε με την προσέγγιση του εισηγητή όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων καταναλωτών. Έτσι θα τα καταφέρουμε καλύτερα με την τροπολογία, με την τροποποίηση τέλο πάντων της οδηγίας για τις καθολικές υπηρεσίες και τελικά συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης όσον αφορά την ε, σκοπούμενη κωδικοποίηση παρά το ότι γενικά συμφωνούμε με τον εισηγητή έχουν ε, υποβληθεί 300 τροπολογίες και εγώ ως σκιώδες του ΕΛΚ. Έχω υποβάλει 18 τροπολογίες για να βοηθήσω στο να βελτιωθεί το σχέδιο έκθεσης. Τεχνικού χαρακτήρα τροπολογίες έχουμε υποβάλει επίσης που αφορούν τις αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού για τις καθολικές υπηρεσίες. Έχουμε απαλληφθεί κάποιων διατάξεων αιτιολογικών ε, αιτιολογικών παραγράφων ε, κλπ. Γιατί δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται να επαναληφθούν αυτέ οι δύο τάξεις που έχουν σχέση με το δικαίωμα των καταναλωτών. Από την άλλη μεριά όμω, έχουμε υποβάλει κάποιε τροπολογίε για να βελτιώσουμε την αρχική πρόταση. Όσον αφορά την παράγραφο 3 του άρθρου 21, σε αυτό το σημείο διαφωνούμε με τον εισηγητή, γιατί θέλει να διαγράψει όλο το άρθρο. Έχω την τροπολογία 147. Εκεί λέει ότι δεν θα πρέπει να σβήσουμε τη διάταξη που αφορά με τις δυσμενείς διακρίσεις επί τη βάση του τόπου διαμονής και ηθαγένειας ε, θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Επίσης, ελεύθερη, ελεύθερο δικαίωμα, απόλυτο δικαίωμα ελευθερία εγκατάσταση. Ε, αυτά αφορούν τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θεωρούμε ότι αυτέ οι αρχέ πάντοτε αξίζει να προστατεύονται. Και συμφωνούμε ότι το να συγκροτηθεί ένας μηχανισμός για να ρυθμίζεται συγγνώμη λέει συμφωνούμε με το ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός να ρυθμίζει τα της κατανάλωσης. Εάν δεν συνεπάγεται κόστος για τους καταναλωτές. Για το switching. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε μία εργάσιμη. Παρά το ότι είχε πίεση χρόνο έκανε συμβαστικές τροπολογίες ο σύγητης για τα άρθρα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών. Οπότε θα πρέπει και πάλι να εξάρουμε το έργο του εισηγητή. Στις 7 Ιανουαρίου συναντήθηκαν οι σχεδόν εισηγητές, συζητήσαμε τις συμβαστικές προτάσεις και γενικά υπήρξε συνένεση. Τώρα Περιμένουμε πώς και πώς τις προτάσεις, τις συμβαστικές του εισηγητή για τα υπόλοιπα θέματα. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι υπάρχει αυτή η συνένεση και άρα και για τα υπόλοιπα θέματα θα τα βρούμε εν κατακλείδη. Να είναι σίγουρος ο εισηγητής ότι θα συνεργαστεί με του το ΕΛΚΟ τόσο να έχουμε ένα κανονισμό που να προστατεύει τον κατάλληλο και να ε, συμβάλλει στη δημιουργία της ε, ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Ο κύριος Άγκστρομ είναι ο μόνος σκιώδης που παρίσταται. Κύριε Άγκστρομ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς ε, για την πολύ καλή και επικοδομητική δουλειά που κάνατε. Στη συνάντηση σχεδόν εισηγητών ήταν πολύ επικοδομητική η δουλειά που κάναμε. Και όπως αναφέρθηκε βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να επιτευχθεί συνένεση για την πτυχή της προστασίας των καταναλωτών. Πολύ καλή αυτό. Και προσβλέπω ιδιαίτερα φυσικά στη συζήτηση προσβλέπω όσον αφορά την αμεροληψία, την ουδετερότητα όσον αφορά το δίκτυο. Αυτό είναι το θέμα το οποίο πραγματικά μας ενδιαφέρει. Πρέπει να διασφαλίσουμε ιδιαίτερα ότι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες δεν θα έχουν κάποια δυνατότητα δούριου ύπου ή παράθυρο να υπεκφεύγουν και να εξαιρούνται. Το διαδίκτυο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σήμερα για οποιασδήποτε επιχειρήσεις που θέλουν να συναλλάσσονται πανευρωπαϊκά έχει πραγματικά μεγάλη σπουδαιότητα αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε να προστατεύουμε ένα ανοιχτό, <clears throat> καλό λειτουργούν δίκτυο, δίκτυο. Πρέπει να δούμε το τι θα συμβεί και την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πρόεδρος Ελπίζω να μην σας απογοητεύσω, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσει να προχωρήσει η συζήτηση. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή και πρόεδρό μας για την εξαιρετική δουλειά που έκανε μέχρι τώρα. Η ουσιοδέστερη προσέγγιση είναι κάτι που χαιρετίζουμε ιδιαίτερα. Αφενός δηλαδή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ένα ή άλλο σημείο να μπορέσουμε να το θεμελιώσουμε και βελτιώσουμε. Έγινε αυτό και για το θέμα της προστασίας των καταναλωτών αυτό είναι ένα σημείο που θα είχα μια επερώτηση προς τον εισηγητή για την επίτευξη των συμβαστικών αυτών προτάσεων που εξέθεσε. Στον συμβιβασμό γίνεται λόγος για fixed data links, δηλαδή αυτό το οποίο αναμένεται σε ένα ε, ελάχιστο επίπεδο. Αυτό εξετέθη προφορικά πιο πριν. Ερωτώ, τι αναμένουμε τι σημαίνει αυτό το οποίο αναμένεται ως συνήθως ακριβώς. Δηλαδή παίρνουμε ένα μέσο όρο ετήσιο μέσο όρο δεν αποσαφηνίζεται επαρκώς για μένα. Γι' αυτό θα ήθελα πραγματικά τα στοιχεία που αφορούν ε, την ελάχιστη, τα ελάχιστα αυτά επίπεδα στο κείμενο, ώστε να είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών πρέπει να αποσαφηνίζουν ποιο δυναμικό έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να μην ε, επαναλαμβάνεται στη διαφήμιση αυτό το οποίο συμβαίνει μέχρι σήμερα, δηλαδή να μεγιστοποιούν τα πράγματα εναντί των καταναλωτών σε διαφημίσεις, να γνωρίζουμε ποιο είναι στον το διαθέσιμο δυναμικό σε σχέση με τους παρόχους. Διότι αυτό συνδέεται με το ότι οι επιχειρήσεις πάροχοι τηλεπικοινωνιών με βάση τις συμβάσεις που συνάπτουν με τους πελάτες τους συμβατικούς ε, εταίρους τους πρέπει να διασφαλίζουν αυτή την πτυχή ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Αυτό αφορά η δική μου τροπολογία. Αυτή είναι η ερώτηση μου προς τον εισηγητή. Τι σημαίνει το normally available, το ω συνήθως αναμενόμενο διαθέσιμο. Για το δεύτερο σημείο συμφωνώ με τον συνάδελφο Έγκστρομ στα όσα είπε. Είναι σημαντικό πιστεύω. Αν θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα εξειδικευμένων υπηρεσιών, specialized services, ειδικών υπηρεσιών σε σχέση με ένα ανοιχτό, ελεύθερο διαδίκτυο και να δούμε τι μπορεί να επιτευχθεί και τι θα εξαιρείται, να υπάρχει ένας ορισμός για την ουδετερότητα και αμεροληπτία του δικτύου με ε, μη ε, αμφίσιμο τρόπο υπάρχουν κάποιες προτάσεις που δεν αντανακλούν, αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να προσπαθήσουμε στους συμβιβασμούς να καταλήξουμε σε έναν ε, εφικτό προσδιορισμό της ουδετερότητας και αμεροληψίας και προσβλέπω στη δουλειά που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα αυτός ο ορισμός ε, να επιτευχθεί με καλύτερο τρόπο. Διότι είναι σημαντικό να αποσαφηνίσουμε ότι η ουδετερότητα του δικτύου δεν σημαίνει ότι τα πάντα ή τίποτα, δηλαδή επί παντός του επιστητού ή ε, οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να εντάσσεται ή όχι. Πορνογραφία για παράδειγμα σε σχέση με τα παιδιά ή παράνομο περιεχόμενο. Φτάνουμε σε ένα σημείο που λέμε η φυστάμενη νομοθεσία θα πρέπει να δούμε τι θα επιτρέπει και τι όχι. Στα κράτη-μέλη είναι διαφορετικά τα πλαίσια. Αλλά αυτό δεν μπορεί με αυτή την οδηγία να επηρεάζεται και γι' αυτό πρέπει να δούμε, αν ε, εννοούμε σοβαρά τα πράγματα με την πνευματική ιδιοκτησία, copyright, πρέπει σε αυτό το σημείο να μπορούμε να παρεμβαίνουμε με δικαστικές αποφάσεις για παράδειγμα ή και άλλες ε, ε, σαφείς και καθαρές δυνατότητες παρέμβασης από το νομικό πλαίσιο, νομικό επίπεδο σε σχέση με το διαδίκτυο και σε σχέση με την πορνογραφία και τα παιδιά. Για παράδειγμα στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε ανταλλάξει πολλές φορές απόψει και έχουμε συμφωνήσει και επ' αυτού ότι πρέπει να ε, διαγράφονται, να εξαλείφονται από το δίκτυο τέτοια στοιχεία και να υπάρχει μια ανοιχτή τέτοια παρέμβαση στη ροή δεδομένων. Πρέπει να έχουμε μια, ένα σαφή ορισμό που θα δίνει σαφή ε, όρια αυτών των δυνατοτήτων και αυτό είναι το αίτημα που έχω και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Να ληφθεί επαρκώς αυτή η πτυχή υπόψη. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Άλλοι που θα ήθελαν να παρέμβουν, εσείς παρακαλώ. Εξ ονόματος της Ρούζα Τούν εγώ θα παρέμβω. Ναι. Αν... Ακολουθώντας αυτά που είπατε, είναι σαφές ότι οι ορισμοί πρέπει να είναι σαφείς, σαφέστατοι. Συμφωνώ. Υπάρχουν πολλές φορές διατυπώσεις που ακούγονται όμορφες αλλά δεν γνωρίζουμε τι κρύβεται πίσω από αυτές. Έχω καταθέσει και εγώ τροπολογίες ε, για την διαγραφή του κόστους ε, των τελών περιαγωγής, roaming charges. Και αυτό είναι ένα αίτημα που υπάρχει. Οι λύσεις ε, αναμένουμε να δοθούν, προσβλέπουμε στο να εξευρεθούν λύσεις για τους πολίτες που προσδοκούν να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Και ελπίζω ότι θα μπορέσει αυτό να διευθετηθεί λοιπόν όπως πρέπει. Το phasing out όσον αφορά τα πρόσθετα τέλη για την περιαγωγή. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί, πρέπει να είναι προτεραιότητα για μας εδώ. Right. if else... Μάλιστα. Αν δεν θέλει κάποιος να παρέμβει, ζητώ τον, από τον Άντωνι Γουίλεν να παρέμβει και να σχολιάσει. Ίσως έχει και περαιτέρω σύμβουλες να μας δώσει όπως θα του ζητούσα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Λυπούμε ότι πρέπει να πω ότι σε σχέση με την πορεία προς τη Δαμασκό <laughs> μεταξύ Σούμαν και Κοινοβουλίου δεν μπορώ να πω ότι σε σχέση με την ε, συνδιαλλαγή για την οποία έχω προσκληθεί για την αλλαγή κατεύθυνσης ε, και μέσου που προτείνατε Πρόεδρε αλλά σημειώνω με προσοχή τα όσα αναφέρονται και την κίνηση που σημειώθηκε προς ε, αυτή την κατεύθυνση από την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή. Πρέπει να αποφύγουμε φυσικά να αποφύγουμε το να καταλήξουμε να είμαστε αιμονικοί και να έχουμε αιμονές όσον αφορά την ε, γενική αναζήτηση της επίτευξης του γενικότερου στόχου. Να πετύχουμε δηλαδή στο να υπάρχουν κοινοί όροι και προδιαγραφές για τη λειτουργία και τους παρόχους υπηρεσιών στο δίκτυο στην Ευρώπη και κοινού όρους και προϋποθέσεις για την κατανάλωση, για τους καταναλωτές ε, για αυτές τις υπηρεσίες. Έχοντας λοιπόν ε, <clears throat> σημειώσει την ε, μόνιμη προτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη αυτού του στόχου, επιτρέψτε μου να σχολιάσω κάποιες από τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στις συμβαστικές τροπολογίες και τις άλλες τροπολογίες από το Ευρωκοινοβούλιο που φυσικά βρίσκονται υπό άλλο πρίσμα ή άλλη προοπτική αλλά ε, συμμερίζονται τον στόχο, την επίτευξη του στόχου. Πρώτα απ' όλα και δεν θα προσπαθήσω εδώ να αναφερθώ ε, σε κάθε στοιχείο ε, αυτών των προτάσεων. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οποιοδήποτε και να είναι το μέσο ή εργαλείο ή εν πάση περιπτώσει ακόμα περισσότερο αν αυτό είναι το μέσο το οποίο προτιμά ο εισηγητής και τα άλλα μέλη της, Ευρωπαϊ... της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής τότε τα μέσα και τα εργαλεία με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί ενιαία μορφή και με την αναγκαία ελαστικότητα και ευελιξία πρέπει να εξετάσουμε ακόμα περισσότερο και να εστιαστούμε σε αυτό το θέμα ακόμα περισσότερο. Καλωσορίζουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πείρα και την βοήθεια που μπορεί να δοθεί για παράδειγμα σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές για διαφορετικά θέματα που μπορεί να αναφύονται για να υπάρξουν κοινά αποτελέσματα σε αυτό το εγχείρημα. Θεωρούμε ότι πολύ σημαντικός ρόλος πρέπει να καλυφθεί από τα δεσμευτικά μέτρα σε κάποιους τομείς. Δεύτερο, Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω το γεγονός ότι σε αρκετές πτυχές, αν τα είδα και τα κατανόησα σωστά, οι τροπολογίες οι συμβιβαστικές θα ήθελαν να, να εντάξουν ουσιώδη στοιχεία από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίσως όχι με ιδιώσιμους ε, ταυτόσιμους όρους, αλλά στοιχεία ακόμα και τα οποία δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί και όπου με χαρά βλέπουμε ότι αναπτύσσεται μια αυξανόμενη συνένεση. Θέματα δηλαδή επί των οποίων θα θέλαμε να δούμε να εντάσσονται σε ένα εναρμονισμένο εγχείρημα, σε μια εναρμονισμένη δράση ως πλαίσιο. Θα καλωσορίζαμε ιδιαίτερα ακόμα και έχοντας εσείς τονίσει ότι υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν το μήνυμα αν το έλαβα σωστά για το θέμα της δέσμευσης bundling όσον αφορά τις υπηρεσίες από τους παρόχους πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφοροποιούνται οι διάφορες δυνατότητες. Η λογική ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι πολύ λεπτομερείς διατάξεις των υφιστάμενων διατάξεων για την λήξη συμβάσεων Προ προς όφελος των καταναλωτών και του, του ανταγωνισμού θα μπορούσε να α, α, από, να τύχει, ας το πω έτσι, μη υλοποίησης, να μην υλοποιηθεί σωστά αν δεν είχαμε τις, ε, αναγκαίες αυτές προδιαγραφές για τους παρόχους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσυπογράφαμε και θα θέλαμε να το εξετάσουμε περισσότερο μαζί σας κατά το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Εξίσου, με χαρά βλέπουμε περαιτέρω μηνύματα να αποστέλλονται σε σχέση με το γενικότερο ε, θέμα του ελέγχου ε, και της κατανάλωσης Σημειώνουμε επίσης το αίτημα της κυρίας Μπάστος που διατυπώθηκε σε σχέση με αυτό, καθώς επίσης και το θέμα της χρονικής περίοδου για το switching, για την αλλαγή συμβολέων. Επίσης ε, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε το μήνυμα που αποστέλλεται ότι ο πάροχος είναι το ενδεδειγμένο συμβατικό μέλος για την κάλυψη των ε, ε, δομών ή υποδομών που υφίστανται. Για τα θέματα του 1 και του 2 που γνωρίζουμε ότι είναι μια πτυχή του σημερινού καθεστώτος που δημιουργεί και κάποιες δυσκολίες στην εφαρμογή και υλοποίηση Φυσικά καλωσορίζουμε το γενικότερο ενδιαφέρον των μελών της Επιτροπής που έχει μόνιμο χαρακτήρα σε αυτό το θέμα. Είναι μονιμότερο στοιχείο θα το κατανοήσετε. Είμαστε κάπως επιφυλακτικοί σε μια διαδικασία που συνειδητά προσπαθήσαμε να ενταχθούμε σε θέματα που θα επιταχύνουν την επίτευξη του στόχου της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και τις προβλέψεις και διατάξεις για τους καταναλωτές. Είμαστε διστακτικοί στο να επεκτείνουμε αυτό το ίχνος, αυτό την εμβέλεια αυτής της πρότασης χωρίς να έχουμε μελέτη επιπτώσεων προηγούμενα. Και σε σχέση με την εποπτεία και την εποπτική δράση επιτήρησης από πλευράς μας και αυτό σε σχέση με όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τώρα στο θέμα του ανοικτού δικτύου και των εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως είπατε Πρόεδρε, έχετε ακόμα αρκετή δουλειά τις επόμενες ημέρες με τους σκιώδεις εισηγητές για να επιτευχθούν συμβαστικές τροπολογίες ως προς αυτό το θέμα. Θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομος σε αυτό το θέμα. Φυσικά είμαστε στο πλευρό σας για την ανάγκη να υπάρξουν οι σαφέστεροι όροι για την αντιμετώπιση αυτού του αμφίσιμου επίμαχου θέματος. Ακολουθούμε και παρακολουθούμε με τους συναδέλφους μας και σε σχέση με τη συνέχεια μιας μακράς συνεργασίας επί σειρά ετών την προσπάθεια να εξειδικεύσουμε τις σκέψεις μας και τον προβληματισμό μας για να καταλήξουμε σε θετικές προτάσεις όσον αφορά το σχέδιο προτάσεων. Να υπενθυμίσω κάτι αν επιτρέπετε το οποίο προανέφερα επ' αυτού ότι η ανάγκη αναζήτησης για τη σαφήνεια δεν, δεν πρέπει να μας παγιδεύει σε τεχνικού χαρακτήρα έννοιες και θέματα τα οποία τα προσπερνάμε ταχύτατα η εξέλιξη των πραγμάτων, η πρόοδος που σημειώνεται τεχνικά και τεχνολογικά. Δεν είναι όλα καταγραμμένα σε, στις, ε, δέλτους ε, ε, και στο δεκάλογο ας το πω έτσι των θεσφάτων. Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα θέματα που είπατε πρόεδρε και εσείς να επικεντρωθούμε σε κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών των ενιών όπως εξειδικευμένων υπηρεσιών και προσβλέπουμε στο να συνεχίσουμε τη δουλειά μαζί σας επ' αυτού. Ευχαριστώ. Well, thank you for a very constructive response. ευχαριστούμε για αυτήν την επικοδομητικότατη απάντηση. Δεν σας έχω βέβαια πείσει ακόμη για την προσέγγισή μας υπέρ των καταναλωτών. Αλλά θέλω να σας πω ότι οι τροπολογίες μπορεί να φαίνονται υπερβολικές λόγω των πολλών αλλαγών, αλλά οι βασικές τους ιδέες ε, είχαν πρωτοεκφραστεί στην οδηγία για τις καθολικές υπηρεσίες από το 9 ήδη και μιλούν ήδη τότε για τις ταχύτητες που προβλέπουν τα συμβόλαια. Και εμεί θελήσαμε να βελτιώσουμε την αρχική πρόταση της Κομισιόν από το 2009. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει καμία διαφωνία ότι πρέπει να βοηθηθούν οι καταναλωτές. Θέλουμε απλώς να δούμε πώς θα συνεχίσουμε το δρόμο που άνοιξε από το 9 και θέλουμε να πιέσουμε τους προμηθευτές και τους ρυθμιστές για βελτίωση της χορήγησης των υπηρεσιών αντί για ολόκληρη νέα οδηγία και εναρμόνιση που κατ' εμάς θα ήταν αρνητική για τους καταναλωτές. Λυπάμαι που το ξαναλέω, αλλά εδώ παραμένουμε σε διαφωνία. Βλέπετε όμως ότι το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να κινηθεί προς την κατεύθυνση που σας λέω και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει στάση. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς τελικά θα υπερισχύσουμε γιατί συμφωνούν περισσότερο η πρότασή μας με το κλίμα των καιρών. Λοιπόν, ο κανονισμός αυτός ε, πρέπει να συνδυαστεί με τον κανονισμό που θα αφορά τις ε, συνδυασμένες υπηρεσίες και με τη δυνατότητα να διακόπτονται τα συμβόλαια. Λοιπόν, τώρα να απαντήσω σε μερικά άλλα θέματα που έδειξαν οι συνάδελφοι. Χαίρομαι γιατί η Κομισιόν μας μίλησε και για το θέμα της τεχνολογικής ουδετερότητας ιδιαίτερα ως προς τον κανονισμό για την ανοιχτή πρόσβαση στο ίντερνετ. Δεν ξέρω αν χρειάζεται όντως οριστός τέτοιος κανονισμός, αλλά θα το προσέξουμε ιδιαίτερα. Για την κυρία Χένσελ φοβάμαι ότι διαφωνώ, διότι αν συμπεριλάβουμε όλα όσα μας πρότειναν και όλες τις διατυπώσεις, θα καταλήξουμε σε έναν ορισμό τελείως δυσνόητο και νομικά αβέβαιο. επανέρχομαι σε αυτό που είπα. Πρέπει να κινηθούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση για να επικεντρωθούμε στα κύρια αιτήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η ουδετερότητα, η τεχνολογική ουδετερότητα δεν έχει καθοριστεί γιατί δεν συμφωνεί κανείς περί του τι ακριβώς σημαίνει. Είναι ήδη δύσκολο ως αρχή και ο κανονισμός υποτίθεται ότι θα λύσει αυτό ακριβώς το θέμα. Άρα δική μας δουλειά είναι εδώ να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα και να καταλήξουμε σε διατυπώσεις που να μπορούν να καθοδηγήσουν τους εθνικούς ρυθμιστές ώστε και στην εθνική νομοθεσία να μην εισαχθούν νέες έννοιες γιατί έτσι δεν θα μπορούν οι επενδυτές στις τηλεπικοινωνίες και οι προμηθευτές να αντιμετωπίσουν τέτοιες αβέβαιες καταστάσεις και καθεστώτα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα δείτε θετικά τις ιδέες και την προσέγγιση μου. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα τη δεχτούν όλοι βέβαια, αλλά ως βάση συζήτησης. Οτιδήποτε όμως προσθέσουμε στον κυρίω ορισμό πρέπει να έχει κάποια σημασία, κάποια υπεραξία ως προς τη δυνατότητα των εθνικών ρυθμιστών να καθοδηγηθούν. Θα περιμένω λοιπόν τις απαντήσεις σας την επόμενη εβδομάδα. Για τα άλλα θέματα τώρα, κυρία Μπάστος. Τα απάντησα νομίζω όλα όσα έθιξε. Όσο για τη μέτρηση της ταχύτητας. Αυτό είναι δύσκολο αν θέλουμε λιτή διατύπωση. Ευχαριστώ την προσοχή της κυρίας Βαν Χέινς στις συμβιβαστικές τροπολογίες στη σελίδα 17 γιατί εκεί θα δει ότι στο καινούριο 3α, 3α νέο απαιτούνται γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της ταχύτητας των επικοινωνιών στο Ιντερνετ. και ίσως και ένας μηχανισμός πιστοποίησης ποιότητας. Βέβαια δεν μπορούμε εδώ να αναφέρουμε συγκεκριμένους αριθμούς, ούτε και σε παράρτημα, γιατί αυτά θα αλλάζουν συνέχεια. Και ιδίως όταν μιλάμε για κινητή ίντερνετ ε, σύνδεση, εκεί υπάρχουν ακόμη περισσότερες αλλαγές και διακυμάνσεις ανάλογα με την τοποθεσία όπου βρίσκεται κανείς τη γεωγραφία του χώρου κατά πόσον ε, βρισκόμαστε στην πρωτοχρονιά όπου υπάρχουν πάρα πολλές ταυτόχρονες συνδέσεις κλπ. κλπ. Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποια σαφή βάση για να τα πούμε όλα αυτά και η σαφέστερη είναι ποια είναι η κανονική ταχύτητα, η μέση ταχύτητα. και ποιες είναι οι ελάχιστες ταχύτητες που μπορεί κανείς να αναμένει σε περιόδους μεγάλου φόρτου. Αυτά είναι τα βασικότερα νομίζω. Και ήδη οι διάφοροι ρυθμιστές έχουν αρχίσει να τα βλέπουν όλα αυτά και καμιά φορά ε, υπήρξαν και μηνύσεις κατά προμηθευτών που δεν χορηγούσαν την, την υπεσχημένη ταχύτητα. Στην πληροφόρηση που πρέπει να έχει κανείς πριν υπογράψει λοιπόν το συμβόλαιο, πρέπει να υπάρχει και μία επαλήθευση στη συνέχεια, ώστε όσοι υπογράφουν ένα συμβόλαιο να γνωρίζουν ακριβώς τι να περιμένουν τα καλύψαμε όλα αυτά νομίζω λέγοντας ότι τον πιο λεπτομερή ορισμό θα τον κάνουμε αργότερα. Αν είναι απαραίτητο μπορούμε να ξαναδούμε την αιτιολογική έκθεση και θα δούμε τι λέει εκεί η Κομισιόν για να δούμε αν μπορούμε να το βάλουμε και αυτό στο συμβιβασμό. Λοιπόν, Εκτός αν έχει κανείς τίποτε άλλο να προσθέσει, σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξανασυναντηθούμε για τα θέματα της πρόσβασης στο Ιντερνετ και θα τα εγκρίνουμε αυτά τέλη Ιανουαρίου ώστε στην Επιτροπή Βιομηχανίας να εξεταστεί τέλη Φεβρουαρίου. Δεν νομίζω ότι θα ξανασυζητήσουμε δημόσια εδώ τις συμβιβαστικές. Αν όμως χρειαστεί θα πρέπει να γίνει την παραμονή της ψηφοφορίας. Ελπίζω μέχρι τότε όμως να έχουν τελειώσει όλα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το τελευταίο σημερινό μας θέμα, το Solvit. Solvit, Molvit. Ο κύριος Λούκγκαρντ είναι εδώ. Έρχεται λέει από το αεροδρόμιο. Στις 11 και 20 είχε πει ότι θα έρθει και είναι ήδη 11 και 19.30. Δεν τον βλέπουμε. Κανείς δεν τον βλέπει. Μήπως να του μιλήσουμε στο κινητό του. Γιατί αν αργήσει πολύ τότε θα ανοίξει η συνεδρίαση. Να περιμένουμε πέντε λεπτά λέτε. Να περιμένουμε τουλάχιστον ως τις 11.30. Οι συντονιστές κανονικά πρέπει να διασφαλίζουν ότι έρχονται οι συγχυτές. Εν καιρός, γιατί είναι αγενές τελικά. Και αν δεν έχει έρθει ο κύριος Λόκεγκαρντ, θα δούμε τι θα κάνουμε με την έκθεσή του.

Uh, right, uh, ladies and gentlemen, I um, um, ορίζουμε τον εισηγητή που από την Ταϊβάν, Ταϊβάν έφτασε κατευθείαν σε εμά είναι ενδιαφέρον αυτό και από το αεροδρόμιο κατευθείαν εδώ για να παρουσιάσει τις τροπολογίες του στην έκθεσή του ίδιας πρωτοβουλίας για το Solvit και την κυρία Τούν και την ε, παρουσίαση εκπροσώπηση της κυρίας Χάνσλικ. Ε, Καλώς ορίζουμε τους συναδέλφους και εγώ εκπροσωπώ τον συνάδελφο που είναι σκιώδης εισηγητής των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών και οποιονδήποτε άλλο θέλει να παρέμβει. Καλωσορίζουμε και την κυρία Γκρόβεν από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που θα μπορέσει να σχολιάσει και τις τροπολογίε επίσης. Με χαρά καλό τον εισηγητή να λάβει τον λόγο και να μας παρουσιάσει τις απόψεις του για τις 49 τροπολογίες που κατατέθηκαν στην έκθεσή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλή χρονιά σε όλους σας. Και όπως μόλις είπε ο Πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή, αλλά μόλις ήρθα από την Ταϊβάν ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία αυτή και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ταϊβάν πραγματικά χρειάζεται την FTA και εξικετεύουν να τα καταφέρουμε. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι ενώπιόν σας και τις διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον τις 49 τροπολογίες τον σχετικά χαμηλό αριθμό τροπολογιών τον εκλαμβάνω ως ένδειξη ότι η δική μου έκθεση έτυχε μιας προσέγγισης με τέτοιο τρόπο θετικής προσέγγισης που δεν υπήρξε μεγαλύτερη αντίδραση. Υπάρχει και συνένεση για το μήνυμα που αποστέλουμε σε σχέση με την έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε σχέση με την, ε, το σχέδιο έκθεσης ε, του Δεκεμβρίου για το θέμα αυτό υπάρχουν και κάποιες επικαλύψεις στις τροπολογίες και έτσι φυσικά προσπαθώ να καταλήξω σε συμβιβαστικές τροπολογίες μεταξύ άλλων που μπορώ να αναφέρω είναι η συνειδητοποίηση σε σχέση με αυτά τα θέματα ο ρόλος των συλλόγων και ενώσεων επιχειρήσεων Αυτά είναι κάποια από τα θέματα, τα σχετικά θέματα. Για να τηρήσουμε την προώθηση, την όθηση για αυτό το θέμα πρέπει να παραμείνουμε στο χρονοδιάγραμμα με την 23η του μήνα για την ε, έγκριση. Το γραφείο μου θα διανύμει στους σκιώδεις εισηγητές τις συμβαστικές τροπολογίες σήμερα ή αύριο και μπορούμε έτσι την επόμενη εβδομάδα να συζητήσουμε τα θέματα. Αν χρειαστεί μπορούμε να έχουμε και συνάντηση σκιωδών εισηγητών σχετικά θα ήταν μια ιδέα αυτή γι' αυτό. Διαφορετικά μπορούμε και με το ταχυδρομείο ηλεκτρονικά να τα διεκπαιρεώσουμε αυτά. Αυτά έχω να πω αυτή τη στιγμή. Προσβλέπω στα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Τούν, παρακαλώ. μικροφώνου. Ε, Κυρία Χάνσλικ, δυστυχώς, δεν μπορεί να παραστεί. Αλλά μου ζήτησε να σας διαβιβάσω τα εξή. Να σας τα πω στα πολωνικά, γιατί στα πολωνικά μου έστειλε το σημείο μου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι πρόκειται για μια μεγάλη μας επιτυχία, πρέπει να συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο όσον αφορά το Σόλβιτ και θα πρέπει να δούμε το ότι έχουν υποβληθεί πάρα πολλέ τροπολογίε οι οποίε θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση οπότε νομίζω ότι οι τροπολογίε ε, είναι θετικέ, θα πρέπει να βελτιώσουν το σύστημα και θα πρέπει βέβαια να υπάρχει και κατάρτιση ε, των ε, εργαζομένων ή θα πρέπει βέβαια να λάβουν υπόψη το, το, πώς θα βρεθεί ο καλύτερο τρόπο για να βελτιώσουμε το σόλτ. Και Βέβαια, εξαρτάται από το πόσο καταρτισμένοι είναι οι εργαζόμενοι, χρειάζονται και περισσότεροι βέβαια ανθρωπίνοι πόροι στο Σόλβιτ. και χρειάζονται επομένως να γίνουν κάποιες σχετικές επενδύσεις ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη συνεργασία των επιμέρους κέντρων και να συμφωνεί συμφωνία με τις τροπολογίες εκείνες που αφορούν την καλύτερη ενημέρωση πολιτών αλλά και επιχειρήσεων για το Solvit και έχει υποβάλει κάποιες τροπολογίες ε, αλλά και άλλοι ε, συνάδελφοι αλλά <clears throat> έχει υποβάλει τροπολογίες και ο ίδιος ο συγητής. Έχουμε πούμε εδώ τώρα κάποια ζητήματα που αφορούν ε, τα ε, συστήματα ασφαλείας. Επίσης ε, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις από την κύριο Χάνσλικ σε σχέση με κάποιες τροπολογίες που αφορούν την ανταλλαγή των αρίστων πρακτικών, κάποιες άλλες τροπολογίες ε, για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ε, εμπορικών επιμελητηρίων και η κυρία Χάνσλικ ε, σύμφωνη με αυτές τις τροπολογίες. Βεβαίω και θα πρέπει έτσι να γίνεται, να υπάρχει ανταλλαγή, θα πρέπει αυτή η ανταλλαγή να γίνει, να γίνει πιο εντατική, να γίνουν σχετικές επενδύσεις και σε συμφωνεί και με το ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση στο Solvit ε, από τους ε, αναπήρους ή από τους ηλικιωμένους. Επίσης, κ. Χάνσλικ συμφωνεί όσον αφορά την ε, παρακολούθηση της προόδου του Solvit τώρα που θα έχουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τα κράτη-μέλη επίσης θα πρέπει να έχουν κάποιες προθεσμίες στις οποίες να θα διεκπεριώνουν τις διαφορές που ανακύπτουν να δούμε πώς θα έχουμε ενιαία βάση δεδομένων σε όλα τα κέντρα σχολή έτσι ε, να έχουμε ενιαία αντιμετώπιση από τα κράτη-μέλη. Να σας σταθμίσουμε τα υπέρ και τα κατά, να δούμε πως θα έχουμε ένα νομοθέτημα που να βελτιώσει την κατάσταση του δικτύου. Πάντως ε, και έτσι αυτά τα πράγματα λειτουργεί πάρα πολύ καλά το Solvit όπως σήμερα ε, ατύπως λειτουργεί. Άρα γενικότερα συμφωνεί η κυρία Χάνσλικ με τις τροπολογίες και ευχαριστεί τους συναδελφούς που τις υπέβαλαν. ευχαριστω ευχαριστώ και τα μέλη. Οι τροπολογίες αυτές είναι τροπολογίες που μπορώ να εγκρίνω και να υποστηρίξω. Συνεχίζω νομίζω να κινούνται προς την ίδια την κατεύθυνση με τις τροπολογίες του εισηγητή. Αυτό που κάνουμε ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικό και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που θα βρίσκονται στο επίκεντρο των τροπολογιών μας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα μέσα και τα εργαλεία που υφίστανται και να τα χρησιμοποιούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίλυση των προβλημάτων. Πολίτες και επιχειρήσεις λοιπόν έχουν το δικαίωμα να βρίσκουν τις σωστές και δικαιότερες λύσεις με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και πρέπει να γνωρίζουν ποια μέσα έχουν στα χέρια τους ως εργαλεία ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να υποφελούνται από τα προτερήματα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Αυτά είναι κάποια συμπεράσματα κέρια σημασίας που ήθελα να αναφέρω. Πόρους και εργαλεία που αναφέρθηκαν και από τους συναδέλφους. Αυτά τα στοιχεία αναφέρω και στις τροπολογίες και πρέπει να πούμε ότι η χρήση του it ε, ή του it πρέπει να είναι υποφελής. Πρέπει να συμπεριλάβουμε <clears throat> και άτομα με ειδικές ανάγκες ε, και τους ε, ηλικιωμένους. Και μια άλλη πρωτοβουλία που προτείνω είναι ότι το it πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες μας και όπου είναι δυνατόν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και στο, τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Ακόμα και αν η αρμοδιότητα είναι κυριότερα των κρατών μελών. Αλλά πρέπει σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο να εντάσσεται ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες. Ε, δύο πτυχές θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ, δύο στοιχεία. Την παράγραφο 24 όπου ο συντάκτης στοχεύει τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των συγκεκριμένων προτάσεων που διατυπώνονται να διαγραφεί. Δεν πρέπει να γίνει δεκτό αυτό πιστεύω εγώ. Μετά στην παράγραφο 25 του σχεδίου της έκθεσης η μέτρηση, η εκτίμηση της πραγματικής πρόοδου που σημειώνεται με το Solvit πρέπει να σταθμιστεί και να δούμε ποια είναι η ε, εμβέλεια αυτής της προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων. Πρέπει να διασφαλίσουμε την επίτευξη των πραγματικών μας στόχων. Αλλά πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να έχουμε και τυπικούς επίσημους στόχους που πρέπει να επιτύχουμε, λαμβάνοντας υπόψη τα επίσημα στοιχεία και ε, συστατικά του Solvit. Να δούμε πώς λειτουργεί το Solvit ακόμα και αν συνεπάγεται διπλή προσπάθεια, διπλή προσπάθεια για να επιτευχθεί. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μηχανισμοί ε, Alternative Dispute Resolution, η εναλλακτική επίλυση διαφορών, εξοδικαστική συμφωνία σε σχέση με διαφορές πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε όλους τους πιθανούς μηχανισμούς και τα εργαλεία σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε πώς οι υφιστάμενοι αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν ώστε να μπορούμε να ε, ωφεληθούμε από την υλοποίηση αυτή στο μέλλον. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Στόχους που τα κράτη σε επίπεδο κρατών μελών για το Solvit πρέπει να επιτευχθούν και υποστηρίζουμε έτσι από κοινού την επίτευξη αυτών των στόχων. Προσβλέπουμε λοιπόν στη συνεργασία με τον εισηγητή και από κοινού με τους άλλους κοιόδης εισηγητές να συνεργαστούμε θετικά για την πρόταση που υποβάλλεται από τον εισηγητή θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και διμερώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αν χρειαστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πιστεύω ότι ηλεκτρονικά μπορούμε να συνεννοηθούμε για αυτά τα θέματα. Πολλές τροπολογίες πιστεύω βελτιώνουν το κείμενο. Ωστόσο, είχα την εντύπωση σε κάποιε τροπολογίες, ε, δυστυχώ ο Ταραμπέλα δεν ε, παρίσταται, ότι δεν συνεισφέρουν υποχρεωτικά σε αυτό το θέμα και δεν εντάσσονται υποχρεωτικά στο θέμα αυτό. Η διαχείριση από πλευρά των κρατών μελών, η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ε, ενθαρρύνει την, ε, τον συντονισμό των περιφερειακών συστημάτων. Δεν είναι έργο του Solvit αυτό. Καλό θα ήταν τώρα να μην ε, λάβουμε τέτοια πρόσθετα βάρη που θα εντάξουμε στο πλαίσιο του Solvit πρέπει να είναι επαρκές τα υφιστάμενα πλαίσια να τηρηθούν και να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει ενώπιόν μας. Σε αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε. Καλύτερα θα ήταν στου, πολίτε πολίτες επ' αυτών να τους ενημερώσουμε. Ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι του Solvit. Παρόμοιες τροπολογίες τέθηκαν και από το Haslick σε σχέση με την ε, τροπολογία 19. Επικέντρωση στα ουσιοδέστερα στοιχεία των στόχων πρέπει να επιτευχθούν. Κατά τα άλλα είναι μια καλή έκθεση και την υποστηρίζω. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, Mrs. ευχαριστούμε. what και εγώ και άλλοι συνάδελφοι που λείπουν που έχουν μιλήσει ε, θεωρούν ότι έχει πάρει σωστή κατεύθυνση η υπόθεση. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Αυτό είναι μια ε, ε, ακόμα ε, πετυχημένη έκθεση που θα διεκπαιριώσουμε και επίσης ο κύριος ε, Φόξ, για λόγους του οποίου σας ομιλώ, είπε ότι κάποιες τροπολογίες κατατείνουν στο να διευρυνθεί το βελληνικές του Σόλβιτ. Είναι θέμα βέβαια εντολή, είναι θέμα ε, δικοδότηση. Some more tasks onto it, uh, for which it's not necessarily equipped. And I think part... Ε, βέβαια, το προσθέσουμε αρμοδιότητες δεν σημαίνει βελτίωση της κατάστασης αναγκαστικά, αλλά θα πρέπει να προκοδοτήσουν τα κρατημέλη ε, το σύστημα πληροφόρησης του Solvit. Το core Solvit να ενισχυθεί, ο πυρήνας του, του, δικτύου. Αυτά γράφει ο κύριος Fox. Ε, Είπαμε προσοχή, να μην ε, απονευρώσουμε την πρότασή μας με υπερβολικούς ε, συμβασμούς. Πρόκειται για μια καθολική υπηρεσία, λέει. Είναι κάτι το οποίο βοηθά την κοινή αγορά. Πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση και εποπτεία. Βοηθούνται. Επίσης, ε, που συσχολούν με την αμοιβαία αναγνώριση των δεξιότητων. Αφορά επίσης το Solvit και βοηθά αγαθά και υπηρεσίες όσον αφορά την εμπορία διακίνησή τους. Πολύ σημαντικό να υπάρχουν σχετικές πληροφορίες. Θα λέει ο κ. και πιστεύω ότι θα είναι ολόψυχα υπέρ της έκθεσης. Θέλει άλλο το λόγο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω ακόμη μια φορά τις ευχαριστίες μας προς τον κύριο Λόκεγκαρτ και τα άλλα μέλη της Επιτροπής σας για την ευρεία στήριξή σας προς το Solvit, όχι μόνο τώρα αλλά και από χρόνια. Επίσης δεχόμαστε τις κριτικές σας, ε, τις επικρίσεις σας ως προς το μόνιμο πρόβλημα για τους πόρους. Είναι και έλλειψη προσωπικού αλλά ίσως και έλλειψη τεχνογνωσίας και επιμόρφωσης του προσωπικού αυτού. Χαιρόμαστε που τα θέτετε αυτά τα θέματα. Άλλο βασικό θέμα, η διαχείριση από το Solvit επιχειρηματικών προβλημάτων. Δεν έχουμε αρκετές επιλύσεις από το Solvit και όσες επιχειρήσεις προσέρχονται και προσφεύγουν στο Solvit δύσκολα λύνονται. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Λόκεγκαρτ για τις επικοδομητικότατες ιδέες του κατά τις διμερί, τα διμερή brainstorming που κάναμε για αυτό το θέμα. Πρέπει νομίζω να δημιουργηθεί περισσότερη διαφάνεια γιατί οι περιπτώσεις των εμπορικές επιπτώσεις έχουν περισσότερο ενδιαφέρον και συμφέρον για τα κράτη-μέλη από ότι οι περιπτώσεις οι υποθέσεις ιδιωτών και γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο να επιληθούν. Συμφωνούμε λοιπόν ότι η έκθεση και οι τροπολογίες κινούνται βασικά προς την ίδια κατεύθυνση με μας τέσσερα σημεία συγκεκριμένα στις τροπολογίες όπου θα ήθελα να επιδειχθεί κάποια φρόνηση γιατί βλέπω διαφορές μεταξύ μας. Πρώτον, η ορατότητα και η δημοσιότητα. Εμείς πιστεύουμε ότι η διαφήμιση του Solvit όπως γίνεται δεν είναι αρκετή. Εμείς θα προτιμούσαμε να προωθήσουμε το U Europe γιατί αυτό είναι ο μηχανισμός που φιλτράρει, που μας δείχνει ότι υπάρχει ένας τρόπος επίλυσης. Αν έχει κάποιος πρόβλημα εμπορικό δεν πρέπει να πάει στο Solvit αλλά στα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών. Επίσης το U Europe δίνει συμβουλές γιατί πολλοί προσφεύγουν στο Solvit ενώ μπορούν τα θέματα να λυθούν αλλού ευκολότερα. Δεν θα θέλαμε λοιπόν να προωθείτε το Solvit ως μοναδική και μεμονωμένη λύση, αλλά να προωθείτε το σύνολο των λύσεων που προτείνει το U Europe. Δεύτερον, η ανάγκη που βλέπουν ορισμένοι για νομοθέτηση του Solvit περαιτέρω το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν με τα κέντρα Solvit και γενικά θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω νομοθεσία. Και ίσως να ήταν αυτό και επικίνδυνο, γιατί από τη στιγμή που μπαίνει κάτι στην νομοθεσία και τα κράτη-μέλη σκληραίνουν τη στάση τους και γίνονται πιο επίσημα και φοβούνται μήπως χρειαστούν πολύ περισσότερες νομικές συμβουλές και διαδικασίες ενώ είναι γνωστό ότι πολλές υποθέσεις δεν πρόκειται να λυθούν σε 10 εβδομάδες, ας πούμε. Το τρίτο θέμα είναι η τροπολογία 37 για την περιφερειοποίηση του Solvit. Θέλουμε περισσότερη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών οργανισμών και Solvit, αλλά μια περιφερειοποίηση φοβούμαστε ότι θα κατέληγε σε κατακαιρματισμό. Τα κέντρα Solvit δεν διαχειρίζονται πάρα πολλές υποθέσεις το καθένα, μερικά μάλιστα 5 με 10 μόνο το χρόνο. Και αν αυτό το κατακαιρματίσουμε και περιφερειακά δεν θα οδηγηθούμε σε καλύτερη εξυπηρέτηση. Υπάρχουν κέντρα Solvit που έχουν μεγάλη εμπειρία επίλυσης διαφορών, έχουν καλύτερες επαφές, είναι θέμα οικονομικής κλίμακας. Και υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος με την περιφερειοποίηση να τα υπονομεύσουμε όλα αυτά. Υπέρ λοιπόν της συνεργασίας αλλά όχι του χωρισμού το Solvit σε περιφερειακά γραφεία. Τέλος υποστηρίζω και αυτά που είπε η κυρία Ρούλε και ο κύριος Χάρμπορ για την ανάγκη να παραμείνουμε επικεντρωμένοι σε συγκεκριμένου στόχους, να μην βάλουμε υπερβολικά πολύ ευρεία εντολή στο Solvit, γιατί δεν θα μπορέσει να επιλύσει πολύ περισσότερες υποθέσεις. Ήδη αν κάνει λύση αυτές που λύνει πιο αποτελεσματικά θα ήταν θετικό. Να παραμείνει δηλαδή γρήγορο και αποτελεσματικό ως επίλυση προβλημάτων για τις επιχειρήσεις και τους παλίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο κ. Λούκεγκορντ να συνοψίσει αν θέλει. Αλλά σας θυμίζω ότι στις 22 Ιανουαρίου και 23 θα ψηφίσουμε, 22 θα συζητήσουμε τις περαιτέρω προτροπολογίες Ναι βέβαια, βέβαια. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι θέλω να σας ευχαριστήσω για όσα είπατε. Γενικά φαίνεται ότι είναι πολύ καλή η προσέγγιση όλων των ομάδων. Θα προσπαθήσω βέβαια να αναλάβω τα περισσότερα από όσα υπόθηκαν ίσως και όλα. Δύσκολο, αλλά ελπίζω να το καταφέρω. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για τις συμβουλές της. Τις έχουμε ξανασυζητήσει σε προηγούμενες μας συναντήσεις βέβαια. Βεβαίως και θα δεχτώ αυτά που είπε για την ορατότητα είναι πολύ σωστά. Επίσης νομίζω για τη διατήρηση της έμφασης εκεί που βρίσκεται σήμερα και για τον μη κατακαιρματισμό, να μην προσθέσουμε και άλλο βάρος στη λειτουργία του. Συζητήσαμε τα νομοθετικά πολλές φορές και για μένα είναι σημαντικό το ξαναλέω η Επιτροπή μας να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα, ηχηρό μήνυμα Και βέβαια στόχος μας δεν είναι να χειροτερέψουμε εδώ τα πράγματα. Θα προσέξουμε λοιπόν ιδιαίτερα τη διατύπωση. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε έναν τρόπο. Αλλά ξαναλέω πολιτικά είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να επωφεληθεί από την παρελθούσα εμπειρία της και να δώσει ένα μήνυμα διεθνώς διεθνώς. Πρέπει βέβαια και τα κράτη-μέλη να πιστούν και τα λέμε πολύ σοβαρά όλα αυτά. Και όταν λέω κράτη-μέλη εννοώ τις επιχειρήσεις. Τώρα, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άκουσα ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε με email, εντάξει, ναι, ωραία. Και νομίζω ότι για τις 22 θα είμαστε έτοιμοι. Ωραία, σας κατευχαριστώ και σας και τους κοιόδης. Πάει και αυτό λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους που συμμετέσχουν και το κοινό μας, το κοινό. Σας υπενθυμίζω ότι January will be on the Wednesday the 22nd. Είπαμε 22 ειπαμε 22 απο τις 9 μέχρι τις 12.30 θα εξετάσουμε τις συμβιβαστικές για διάφορες εκθέσεις και τις προτάσεις μου για τα θέματα της ουδετερότητος καθώς και την έκθεση του κυρίου Λόκεγκαρ, του κυρίου Σφάμπ και το απόγευμα στις 3 ο κύριος Χατζηδάκης θα προσέλθει για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα της ελληνικής Πραεδρίας. Ελπίζω να έρθετε πολύ. Και οι εισηγητές επίσης πρέπει να έρθουν για να του θέσουν ερωτήματα. Και την Πέμπτη θα ψηφίσουμε όλη την ημέρα μόνο θα ψηφοφορίες θα έχουμε. Θα ειδοποιήσουμε αλλά 9 και 4 αντί για 10 για να προλάβουμε και δεν θα χρειαστεί να συνεδριάσουμε απόγευμα εκείνη την ημέρα. Δεν χρειάζεται. Μερικοί θα χαρούν γι' αυτό. Άλλοι όμως όχι. Θα σας δούμε λοιπόν τότε. Καλή χρονιά για όσους δεν το, το είπα. Και θα βρεθούμε στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα όπου και θα χρειαστεί να εγκρίνουμε όλη τη δέσμη των δημοσίων προμηθειών με την οποία ασχολήθηκαν πολλοί. Θα συζητηθεί πέμπτη απόγευμα, την τετάρτη λοιπόν το απόγευμα, τρίτη το απόγευμα στις 3, τρίτη το απόγευμα στις 3 και υπάρχει και η δέσμη του κ. Ροσφόρ για τα καταναλωτικά. Θα σας δω λοιπόν τότε και σας κατευχαριστώ. you can have Ashley's comments